Yeah, that's a sport program and uh, a sport program without costs, huh? so you can show how fit you are and. Έχουμε λοιπόν ένα νέο πρόγραμμα για τον αθλητισμό, το οποίο περιλαμβάνει τη μετακίνηση από τη μία αίθουσα στην άλλη όσο γίνεται πιο γρήγορα. Είναι μια υπηρεσία που παρέχουμε ειδικά για τα μέλη τη Επιτροπή μα. Now we are going to Περνάμε τώρα στα σημεία 15, 16 και 17. Πρόκειται για κοινή συζήτηση σχετικά με την σχέση μας με τη Χιλή και τον εξυγχρονισμό της συμφωνίας. Η συγγήτρια είναι η Μακουλάδα Ροδρίγες και της δίνω κατευθείαν το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ εδώ την πρεσβεία της Χιλιλής και την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης που θα μπορέσουν να απαντήσουν και στις ερωτήσεις μου. Μιλάμε τώρα για δύο συμφωνίες με την ε, Χιλή που περνάνε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις έχουμε από το Σεπτέμβριο. Πρώτον, πρόκειται για μια συμφωνία εμπορική σχετικά με τα βιολογικά προϊόντα και το δεύτερο είναι το πρωτόκολλο τη συμφωνία Σύνδεσης για την προσχώρηση της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, πρόκειται και για συμφωνία ε, σύνδεση με τη Χιλή όσον αφορά τα βιολογικά προϊόντα. Όσον αφορά λοιπόν τα βιολογικά προϊόντα πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω ότι στο Συμβούλιο Γεωργίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε εντολή για να διαπραγματευτεί συμφωνίες που θα διευκολύνουν την εμπορία βιολογικών προϊόντων. Οι διαπραγματεύσει με τη Χιλή έκλεισαν την προηγούμενη εβδομάδα όταν ο Ευρωπαίο Επίτροπο και ο Υπουργό Γεωργία τη Χιλή στι Βρυξέλλε υπέγραψαν την συμφωνία και σύντομα θα μα έρθει και επίσημα στο Κοινοβούλιο. Το κείμενο υπάρχει στο διαδίκτυο και πρόκειται για το αποτέλεσμα μιας ε, πολύ σε λεπτομέρειες ε, δουλειά που έχει γίνει. Διότι θα αναγνωρίσει την πιστοποίηση χιλή για όλα τα προϊόντα τα οποία καλύπτονται από την ευρωπαϊκή, από ευρωπαϊκή ρύθμιση. Επίσης και η Ευρωπαϊκή Ένωση δέχεται τα προϊόντα της χυλής αφού προηγουμένως έχει διαπιστώσει ότι υπάρχει ισότιμο επίπεδο προστασίας, ότι τηρούνται οι προδιαγραφές, επίσης ελέγχου όπως γίνεται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατόπιν όλων αυτών αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην αναγνωρίσει τις προδιαγραφές και την πιστοποίηση για ζωικά προϊόντα τα οποία μπαίνουν στην κατηγορία των βιολογικών. Η Χιλή δεν έχει ρυθμίσει ακόμα την βιολογική της ε, εκτροφή και θα δεχτεί όμως η Χιλή την ευρωπαϊκή πιστοποίηση χωρίς όμως να υπάρχει αμοιβαιότητα. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δέχεται ούτε τις ηχθειοκαλλιέργειες με προέλευση τη Χιλή. Στην έκθεση λέμε ότι για να κρυθεί ένα προϊόν βιολογικό, δεν θα πρέπει να υπάρχουν μέσα συστατικά από τρίτες χώρες για τις οποίες δεν έχει εγκρίνει ισοτιμή Ευρωπαϊκή Ένωση. Δημιουργείται μια κοινή επιτροπή επίσης, η οποία ελέγχει την εφαρμογή και, τον, ε, και ενημερώνει τον κατάλογο των προϊόντων. Και μια άλλη ρήτρα εξασφάλισης είναι ότι οποιαδήποτε από τι δύο πλευρέ μπορεί να πάυσει την ισοτιμία εφόσον διαπιστωθεί ότι η άλλη πλευρά δεν τηρεί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη συμφωνία. Βάσει λοιπόν της πρότασης αυτή, πιστεύω και θεωρώ ότι έτσι καλύπτονται οι πιο υψηλέ προδιαγραφέ της Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως θέλω να εκφράσω κάποιε απόψει εδώ για να τι ακούσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι ερωτήσεις. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, ποια θα είναι η σύνθεση της κοινή αυτής επιτροπής και με ποιο τρόπο θα συμμετέχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει πλήρως να ενημερώνεται και να συμμετέχει σε ό,τι έχει να κάνει με τη συμφωνία αυτή. Δεύτερον, με την έγκριση τη συμφωνία αυτή. Μιλάμε για μια περίοδο τριών ετών. Θέλω λοιπόν να γνωρίζω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να κάνει αξιολόγηση αντικτύπου πριν την εκπνοή της προθεσμίας αυτής, ώστε το Κοινοβούλιο και όλοι εμείς να είμαστε παρκώς ενημερωμένοι για να ξέρουμε κατά πόσο είναι καλό ή όχι να επεκταθεί η συμφωνία αυτή χρονικά ή όχι, να παραταθεί δηλαδή. Έπειτα, η αμοιβαία αναγνώριση των ε, πιστοποίησεων για τα βιολογικά. Υπάρχει κάποια εκστρατεία πληροφόρησης προς τους καταναλωτές και τους παραγωγούς για να ξέρουν πώς μπορούν να επωφεληθούν από αυτή τη νέα πιστοποίηση. Και θα τελειώσω έτσι με τα βιολογικά προϊόντα και έρχομαι τώρα στο πρωτόκολλο της Συμφωνίας Σύνδεσης για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας. Είναι ένα καθαρά τεχνικό θέμα και έχει να κάνει με την υποχρέωση που έχουμε να ληφθεί υπόψη η συμφωνία αυτή, λαμβάνοντας υπόψη επίσης και την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και πρέπει να υπογραφεί επιπλέον πρωτόκολλο ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Χιλή για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση ακριβώς αυτή. Επίσης θέλω να ρωτήσω κάποια πράγματα ακόμα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρώτον, τι μεθοδολογία έχει χρησιμοποιήσει στους υπολογισμούς της. Δεύτερον, τι συνέπειες προβλέπει από την προσαρμογή αυτή για τους Ευρωπαίους παραγωγούς. Και τρίτον, αυτή η τροποποίηση μπορεί να έχει δημοσιονομικές επιπτώσεις, στον προπολογισμό δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τέλος, για να τηρήσω το χρόνο μου, θα μιλήσω για την, για τον εξυγχρονισμό της, ε, του τρίτου πυλώνα της Συμφωνίας Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Χιλής. Ξέρουμε ότι πολύ σύντομα θα ολοκληρωθεί η μελέτη αντικτύπου που θα αποτελέσει και τη βάση προκειμένου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει κατευθυντήρες γραμμές για τις διαπραγματεύσεις. Εμείς επανειλημμένως έχουμε πει ότι πρέπει να υπάρξει εξυγχρονισμός της συμφωνίας που ισχύει τώρα και για το περιεχόμενο, αυτό το μήνα θα υποβάλω μία έκθεση που ελπίζω να στηρίξουν όλοι. Έτσι κι αλλιώς είμαι σαφώς υπέρ του εξυγχρονισμού. Την προηγούμενη εβδομάδα πάντως ήμουν άμα τον Υφυπουργό Εξωτερικών της Χιλής και πήγα και στο Σαντιάγο και είδε και την πρόεδρο Βασιλέρ και κατάλαβα ότι μία τέτοια αλλαγή προδευτική είναι κάτι το αφικτό και για τις δύο πλευρές και μπορούμε να το πετύχουμε. Τέλος, στη συμφωνία αυτή θέλω να πω στην Επιτροπή ταξής. Ποιες είναι οι προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη διαπραγμάτευση αυτή και τι επίπεδο φιλοδοξίας περιμένει να πετύχει όσον αφορά την βιώσιμη ανάπτυξη. Υπάρχει περίπτωση να συμπεριληφθεί επίσης ιδιαίτερο κεφάλαιο για την ισότητα των δύο φύλων. Η τεχνική διαπραγμάτευση έχει ολοκληρωθεί στην Ουρουάη. Πρέπει να προσθεθεί πιστεύω ένα τέτοιο κεφάλαιο. Δεν είναι δυνατόν να είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή που μένει πίσω. Δεύτερον, πώς θα εξασφαλίσετε την μέγιστη διαφάνεια στις διαπραγματεύσεις και την ε, καλύτερη συμμετοχή της κοινωνίας των ε, πολιτών και του Κοινοβουλίου. Στα Ισπανικά που είναι επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Χιλής θα υπάρχουν ε, τα κείμενα της συμφωνίας. Και τέλος, προς την πρεσβεία της Χιλής, θέλω να ρωτήσω το εξή. Σε τι βαθμό έχετε δεσμευτεί στο IS. Ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε το λόγο, Πρόεδρε. Κάποιες απλές ερωτήσεις, θα δώσω τώρα το λόγο στους κοιόδης εισηγητές. Ο κύριος Μάτο από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους τους παρόντες που βρίσκονται εδώ. Πολλές είναι οι ερωτήσεις της εισηγήτριας. Δεν θα τις επαναλάβω. Τι να σας πω, είμαι μοιρασμένο όπως λέμε στην Ισπανία. Πηγαίνω προς τη μη και προς την άλλη κατεύθυνση. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα ο στόχος της συμφωνίας όσον αφορά τα βιολογικά προϊόντα φυσικά και είναι πολύ σωστός και ευπρόσδεκτος. Όμως υπάρχουν κάποια ζητήματα εδώ που νομίζω βάζουν πολύ και πρέπει να τα λύσουμε εδώ. Γιατί αφενός μεν συμφωνώ και εγώ ότι είναι καλή η συμφωνία, δεν υπάρχει αμφιβολία, πρέπει να προστατεύσουμε, να δώσουμε όθηση στα εθελοντικά προϊόντα κτλ. Δεύτερον όμω, είμαστε σε μια κατάσταση όπου τώρα ακολουθούμε δύο παράλληλες διαδικασίες, οι οποίες συγκρούνται μεταξύ του μερικέ φορέ. Γιατί εγκρίνουμε από τη μια την συμφωνία την εμπορική και από την άλλη Έχουμε τριμερείς διαλόγους για το εμπόριο ορισμένων συγκεκριμένων προϊόντων γεωργικών, βιολογικών, με σημαντικές συζητήσεις που γίνονται. Είναι αλήθεια, όλοι πιστεύουν στην ισοτιμία και πιστεύουν ότι είναι κάτι καλό. Από την άλλη όμως έχουμε πολύ περισσότερα πράγματα για να πετύχουμε αυτή την ισοτιμία. Στηρίζω λοιπόν, όπως και πολλοί από τους ε, γεωργούς μας, την ταυτότητα, γιατί ξέρετε υπάρχουν προϊόντα όπου η ισοτιμία αυτή δεν είναι πραγματική. Είναι προέλευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν απαγορεύονται σε άλλες χώρες, στην Χιλή για παράδειγμα, Οπότε πρέπει να δούμε ποια είναι τα φυτογενομικά προϊόντα τα οποία γίνονται αποδεκτά. Δηλαδή, την ταμπέλα βιολογικό προϊόν την έχουν προϊόντα τα οποία περνάνε από εντελώ διαφορετική μεταχείριση. Μπορεί να είναι ένα προϊόν που απαγορεύεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί δεν θεωρείται ασφαλές και να επιτρέπεται στην χιλή. Οπότε αυτή η ισοτιμία δεν στέκει. Καλό θα ήταν, εν πάση Να δούμε και την περίοδο. Πέντε χρόνια, πέντε χρόνια, συν πέντε χρόνια. Φοβάμαι ότι έτσι κρατάει υπερβολικά ο χρόνος για να πετύχουμε την ισοτιμία. Δεν είναι αυτό που θέλουμε. Οπότε διαφωνώ με μια τέτοια μεγάλη προθεσμία και για την μπανάνα υπάρχει αυτό το ζήτημα. Πρέπει να είμαστε λοιπόν πολύ προσεκτικοί και να ξέρω εσείς πώς το βλέπετε. Δηλαδή δεν βλέπετε κι εσείς μειονεκτήματα αν υπάρξει τέτοια παράταση. Και κάτι άλλο που μου απασχολεί πολύ είναι οι ακροάσεις της Γενικής Διεύθυνσης ε, ΣΑΝΤΕ που εκεί αναφέρθηκαν προβλήματα που δεν έχουν λυθεί. Οπότε πώς το βλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τον έλεγχο της πιστοποίησης προέλευσης, είναι το ένα. Και το σύστημα ανείχνευσης προέλευσης. Δεν ξέρω, ρωτάω. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να μας δώσει την εγγύηση ότι τέτοια προβλήματα δεν θα εμφανιστούν και πάλι για τη συγκεκριμένη αυτή συμφωνία με τη Χιλή. Και γενικότερα σε συμφωνίες με τρίτες χώρες. Τέλος, πιστεύω ότι είναι καλή η συμφωνία, καλά κάνουμε και την έχουμε, αλλά προσοχή γιατί μπορεί να έχει και αρνητικές επιπτώσεις στα δικά μας προϊόντα. Ευχαριστώ πολύ για το ECR, Αμάμα Κλάρκεν. Ευχαριστώ. Η Χιλή ήταν η πρώτη χώρα τη Λατινική Αμερική που υπέγραψε Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών το 2002 με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν μια νέα γενιά τέτοιων συμφωνιών περιλάμβαναν έναν εμπορικό πυλώνα αλλά και πολιτικό διάλογο και ευρύ φάσμα συνεργασίας που συμπεριλάμβανε επίσης και την ανάπτυξη. Αυτά αύξησαν υπερβολικά, ε, πάρα πολύ το διμερές εμπόριο, όχι μόνο με τη Χιλή. Άνοιξαν τις ε, πόρτες ε, για τη συνεργασία και σε άλλους τομείς, την αλληλεία, την ασφάλεια των τροφίμων, αλλά είναι σαφές ότι το 2017 ε, πλέον μια τέτοια συμφωνία πρέπει να είναι εξυγχρονισμένη για να αντιστοιχεί και να ανταποκρίνεται στις πολιτικές εξελίξεις, στις επιχειρηματικές ανάγκες αμφότερων των πλευρών. Θα πρέπει να είναι πιο φιλόδοξη μια τέτοια συμφωνία και να ε, εκπληρώνει τις ε, μεγάλες προσδοκίες που έχουμε και οι δύο πλευρές. Πρέπει να περιλαμβάνει μια πιο ολοκληρωμένη οργάνωση του εμπορικού πυλώνα και σε πολλούς τομείς η φιλοδοξία της σημερινής ε, συμφωνίας σύνδεσης θα μπορούσε να ενταθεί. Για μας θα θέλαμε να δούμε πρόοδο στο ECR στις δημόσιες συμβάσεις ε, με περαιτέρω δεσμεύσεις αλλά θέλουμε να συμπεριληφθεί και ένα επενδυτικό κεφάλαιο στην συμφωνία σύνδεσης που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Θα θέλαμε να προωθηθεί η ρυθμιστική συνεργασία και οι πρακτικές και να μειωθούν οι διαφορές μέσω της διευκόλυνσης νέων κοινών ε, πρωτοβουλειών για αριθμιστικά ζητήματα. Θέλουμε να συμπεριληφθεί και ένα κεφάλαιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Στη νέα εξυγχρονισμένη συμφωνία φυσικά. Και θέλουμε να δούμε και άλλα στοιχεία όπως την αμοιβαία προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για τα κρασιά. Εμεί στο ECR ελπίζουμε ότι οι συζητήσει εξυγχρονισμού αυτή τη συμφωνία σύνδεση θα ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατόν. αυτή τη στιγμή έχουμε επαρκή πολιτική υποστήριξη ε, και ε, δυναμικότητα για μια νέα συμφωνία. Η ερώτηση που θέλω να κάνω στην Κομισιόν αφορά την εκτίμηση αντικτύπου που πρόκειται να δημοσιευτεί μαζί με τις διαπραγματευτικές οδηγίες ελπίζουμε τον Ιούνιο. Μπορείτε να μας διαφωτίσετε λίγο. Η εκτίμηση αντικτύπου έγινε σε τομείς που αναμένεται αύξηση του εμπορίου και ποιοι ε, νέοι επιχειρηματικοί τομεί θα συμπεριληφθούν και πώ θα επηρεάσει αυτό τι μικρομεσαίες επιχειρήσει. Πιο συγκεκριμένα τώρα όσον αφορά το εμπόριο των βιολογικών προϊόντων και τη συμφωνία που μόλις ε, ε, έχει συναυθεί, μπορείτε να μας εξηγήσετε πώς συνδέεται με αυτή τη συμφωνία και την επικείμενη έναρξη του νέου εξυγχρονισμού του εμπορικού πυλώνα στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων αυτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Ντίτερ, για το Άλντε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ναι, η Χιλή είναι ανοιχτή η οικονομία και αν εξετάσουμε τα δεδομένα των τελευταίων ετών είναι σαφές ότι η παρούσα συμφωνία ελεύθερου εμπορίου ήταν ωφέλιμη κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας ε, για την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, τις επιχειρήσεις της και τα κράτη-μέλη της. Είναι όμως πια ξεπερασμένη και γι' αυτό επικροτώ αυτή την προσπάθεια εξυγχρονισμού για να περάσουμε σε νέα διάσταση στις σχέσεις μας με τη Χιλή. Θα πρέπει να πετύχουμε μια φιλόδοξη και ολοκληρωμένη συμφωνία. Υπάρχει σημαντικό περιθώριο βελτίωση στι εμπορικέ μα σχέσει, για παράδειγμα όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά. Ακούμε συχνά από τις επιχειρήσεις ε, ότι πρέπει να εξετάσουμε το θέμα. Επίσης, γεωργικά προϊόντα, υπηρεσίες, που είναι κλειδί στα, στις νέες ε, συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου. Επίσης, ε, το, το SPS ε, και οι δημόσιες συμβάσεις που είναι κάτι για το οποίο θα πρέπει να ασκήσει πίεση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης θα πρέπει να επιδιώξουμε να υπάρχει κεφάλαιο για τις επενδύσεις και θέλουμε επίσης ένα φιλόδοξο κεφάλαιο για τα δικαιώματα διανοητικής διοκτησίας ε, καθώς ε, και για τα γεωργικά προϊόντα. Γενικά είναι πολλά που μπορούμε να πετύχουμε. Υπάρχει καλή βούληση και από τις δύο πλευρές ε, και νομίζω ότι και υπό τις παρούσες συνθήκες είναι πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει να ασκεί πίεση για την απελευθέρωση του εμπορίου. Ελπίζω το Συμβούλιο σύντομα να μπορέσει να υιοθετήσει την εντολή και να ξεκινήσουμε φέτος τις διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν υπάρχει άλλο σκιώδη εισηγητή στην αίθουσα. Νομίζω όμω ότι ο, ο κύριος Σόλτς θα μιλήσει εκ μέρου ε, τη σκιώδης εισηγήτρια ε, τη ομάδα του. Ε, ναι, πολύ σωστά κύριε Πρόεδρε, η Ελεονόρα Φορέντσα μου ζήτησε να μεταφέρω τι θέσει τη. Δυστυχώ και εκείνη δεν μπορεί να είναι παρούσα σήμερα, αλλά θα Ήθελε να τονίσουμε ότι ήδη το 2003 η συμφωνία με την Χιλή παρουσίαζε κάποιες λήψεις ε, που είχαμε επισημάνει ήδη τότε, ιδιαίτερα το θέμα των κοινωνικών δικαιωμάτων. Καθότι η ισχύουσα συμφωνία καλύπτει το 96% του εμπορίου Ευρωπαϊκής Ένωσης και Χιλής, ε, κάθε εξυγχρονισμός του πυλώνα θα πρέπει να ε, περιέχει κεφάλαιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη, προστασία του περιβάλλοντος και τα δικαιώματα των ε, ηθαγενών, ιδιαίτερα του πληθυσμού Μαπούτσι. Ενθαρρύνεται η εμπορική δραστηριότητα των πολυεθνικών εταιριών ε, και έτσι υπάρχει η ψηλή εκμετάλλευση των ε, φυσικών πόρων. Η Χιλή δεν ήταν σε θέση να προστατεύσει ικανοποιητικά το περιβάλλον ε, και η συμφωνία ενίσχυσε την τάση αυτή. Ε, θέλουμε προστασία του οικοσυστήματος ε, και προστασία της βιοπικιλότητας. Αυτά είναι απλά κάποια παραδείγματα θεμάτων που θα πρέπει να βελτιωθούν στην συμφωνία. Από εδώ θα πρέπει να ξεκινήσει ο εξυγχρονισμό. Θα πρέπει να επενδύσουμε σε ένα ισχυρό πλαίσιο, το οποίο να περιέχει ρήτρε ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων εφαρμόσιμες και να ε, διασφαλίζεται η πρόσβαση σε ένδικα μέσα για τα θύματα. Από το 1973 και μετά η κυβέρνηση της ε, Χίλης ε, δεν ήταν σε θέση να ρυθμίσει θέματα όπως είναι οι δασμοί, οι δημόσιες ε, συμβάσεις και οι επενδύσεις, θέματα που παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην προστασία των δικαιωμάτων σε τροφή, εκπαίδευση κλπ. Θα πρέπει λοιπόν οι διατάξεις για πρόσβαση στην αγορά να λάβουν υπόψη αυτό το γεγονός. Τέλος, όσον αφορά την ρήτρα επενδύσεως, επενδύσεων, θα πρέπει να ε, υπάρχει ε, ένα πλήρες δικαστικό σύστημα που, μπορεί, να μπορεί να χειριστεί πρόσφυγες και να υπάρχει και ένα κεφάλαιο για τις ε, ξένες επενδύσεις ε, και να διασφαλίζεται η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γι' αυτό είμαστε κατά της συμπερίληψης ε, οποιοδήποτε μηχανισμού τύπου ISDS. Όσον αφορά τα βιολογικά προϊόντα και τη συμφωνία αυτή, ναι, μας ανησυχεί το θέμα της ισοδυναμίας διότι αυτό σημαίνει ότι δεν εφαρμόζονται οι ίδιοι αυστηροί κανόνες που εφαρμόζουν οι παραγωγή εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό οδηγεί σε στρέβλωση του ανταγωνισμού. Είναι υψή της σημασίας για τους μικρούς βιολογικούς παραγωγούς και από τις δύο πλευρές του ωκεανού και είναι σημαντικό και για τους καταναλωτές στην Ευρώπη να μπορούν να κάνουν τη διάκριση ανάμεσα στα ευρωπαϊκά βιολογικά προϊόντα και τα προϊόντα που έχουν παραχθεί υπό διαφορετική σειρά κανόνων. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό που είπατε για το ISDS με εξέπληξε. Έχω την τιμή τώρα να δώσω το λόγο στην πρέσβη Φερνάντες. Ε, έχετε το λόγο, παρακαλώ. Μικρόφωνο δεν έχει ο μιλητής. Muchas gracias. Ya, ya, ya. Muchas gracias. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι. Πρώτα απ' όλα, σας ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να απευθυνθώ εδώ στην Επιτροπή Ιντα μια πολύ σημαντική στιγμή στη σχέση της Χιλής με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εγώ αρχίζω τη θητεία μου εδώ στις Βρυξέλλες και πρέπει να σας πω ότι βρίσκω ότι είναι πάρα πολύ θετικές οι σχέσεις της Χιλής με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Συμφωνία Σύνδεσης του 2002 που άρχισε να ισχύει το Φεβρουάριο του 2003 λειτουργήσε παραδειγματικά τόσο το πολιτικό σκέλος όσο και το εμπορικό σκέλος της συμφωνίας αυτής έτσι. Οι εμπορικές σχέσεις πολλαπλασιάστηκαν επί τρία από τότε που άρχισε να ισχύει η συμφωνία αυτή. Συγχρόνως προχωρούμε και σε άλλα θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Μετά από μια μακρά περίοδο διαπραγματεύσεων, η συμφωνία που λαμβάνει υπόψη στην προσχώρηση της Δημοκρατίας ε, της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα εγκριθεί πολύ σύντομα. Έπειτα, η συμφωνία σχετικά με το εμπόριο βιολογικών προϊόντων εγκρίθηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι η πρώτη αυτού του είδους που υπογράφηκε μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τρίτης Χώρας που επιτρέπει στη Χιλή υπό ίσης όρης να μπορεί να έχει προσχώρηση σε μια τόσο σημαντική, την πιο σημαντική βασικά αγορά του κόσμου. Και αυτό με αμοιβαιότητα ανάμεσα στην Χιλή και τις 28 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις πιστοποίησεις βιολογικών προϊόντων. Η έλεγχοι λοιπόν και τα προϊόντα τα οποία έχουν ελεγχθεί και πιστοποιηθεί στην Χιλή μπορούν να περάσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και Τούμπαλιν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για την γεωργία της χώρας μου. Είναι μια ακόμα απόδειξη της δέσμευσή μας υπέρ του βιώσιμου εμπορίου και της βιώσιμης ανάπτυξης. Προχωρούμε βέβαια και στις συζητήσεις για, την, για τον εξυγχρονισμό του τρίτου πυλώνα της Συμφωνίας Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Χιλής, κάτι το οποίο επεσήμανε και η ίδια πρόεδρος Μπασελέρ. Θέλω να υποφεληθώ από αυτή την ευκαιρία για να σας ευχαριστήσω για τη μόνιμη στήριξη που είχαμε από τη δικιά σας Επιτροπή και κυρίως από την εισηγήτρια, την κυρία Μακουλάδα Ροντρίγκες Πινιέρο Φερνάντες, που προχώρησε και στις συνονίσεις με το Συμβούλιο. Και όταν λέω στήριξη, ενώ πλήρη στήριξη, γιατί πάντα την είχαμε από την Επιτροπή σας και από την βουλευτή Ροντρίγε Σπινιέρη, η οποία βοηθάει να εμπλουτιστεί η συζήτηση και να μπορέσουμε να οργανώσουμε καλύτερα τη συνέχεια. Θέλω επίσης να πω ότι συμφωνήσαμε με τις διάφορες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου ε, ότι θα προχωρήσουμε σε, μια, σε ένα φιλόδοξο εξυγχρονισμό δεν υπάρχουν θέματα τα οποία αποκλείονται από τις διαπραγματεύσεις. Γι' αυτό θέλω να πω ότι προβλέπεται και η ένταξη ενός κεφαλαίου ειδικού για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Επαναλαμβάνω τη δέσμευση που έχει αναλάβει η χώρα μου για την πρόθεση των σχέσεων πολιτικών και εμπορικών με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσα από τέτοια συμφωνίες και αυτή που συζητούμε τώρα, όλοι έχουμε να κερδίσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Τέλεια, ευχαριστούμε πολύ και θα μείνουμε σε επαφή για όλα αυτά. Ευχαριστούμε. Να καλέσω τώρα την Κομισιόν και να την παρακαλέσω να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομη, διότι υπήρξαν πολλές ερωτήσεις. Μαζί μας είναι ο κύριος Γιώργενσεν, τμήματάρχης για τη Λατινική Αμερική. Ξανά και η κυρία Έλενα Βανρίτσι από την Γενική Διευθυνσή Γεωργίας. Κύριε Γιώργενσεν. Be... Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο το δυνατόν πιο σύντομος. Ε, ως απάντηση στις ερωτήσεις, πρώτα απ' όλα όσον αφορά το πρωτόκολλο, η μεθοδολογία που χρησιμοποιήσαμε βασίζεται σε γεγονότα είναι αυτή που χρησιμοποιούμε με όλους τους εμπορικούς μας εταίρους και οι συζητήσεις με τη Χιλή ήταν αρκετά εύκολες. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο και χρησιμοποιούμε την ίδια μέθοδο που βασίζεται σε γεγονότα και είναι και αντικειμενική, όπως αυτή που χρησιμοποιήσαμε τις άλλες δύο φορές που είχαμε την ίδια άσκηση με τη Χιλή. Έξω και το αποτέλεσμα. μια κάποια προσαρμογή της ε, δασμολογικής ποσόστοσης για το χείριο που προσφέρουμε στη Χιλή ε, ε, χίλιοι τόνοι παραπάνω το χρόνο και αυτό προστίθεται στις υπόλοιπες αλλαγές που συμπεριλάβαμε σε αυτό το πρωτόκολλο σε σχέση για παράδειγμα με τα πιστοποιητικά τα συγκεκριμένα προγράμματα χώρας για τις υπηρεσίες για τις δημόσιες συμβάσεις, όλα είναι γνώστα. Έχετε δει τα αποτελέσματα και τη μεθοδολογία αυτή και στις υπόλοιπες νομοθετικές πράξεις που έχουν περάσει στο πλαίσιο αυτό ε, για τη Βραζιλία. Ποιες θα είναι οι δημοσιονομικές επιπτώσεις είτε καμία, διότι ουσιαστικά δεν θα υπάρξει καμία αύξηση των ε, αδασμολόγητων ε, εξαγωγών ε, χείρου κρέατος προς τη Χιλή, διότι σήμερα η ποσόστος χείριου κρέατος για τη Χιλή, δηλαδή τα δικαιώματα που έχει η Χιλή για εξαγωγή χείριου κρέατος προς την Ευρώπη δεν τα έχει εκπληρώσει, οπότε μπορεί να συμβεθεί μια μικρή απώλεια μηδενική ή αμελητέα όσον αφορά την επιρροή στα ευρωπαϊκά προϊόντα. Οι κρατικές επιχείρησεις φυσικά θα έχουν περισσότερες δυνατότητες εξαγωγικές. Τώρα κάποια σχολεία για την ε, εξυγχρονισμό. Ποιες είναι οι προτεραιότητες της Κομισιόν. Θα μπορούσα να σας περιγράφω για ώρες. Ε, αν δείτε τις πρόσφατες συμφωνίες μας, ε, τη ΣΥΤΑ ή το έγγραφο διερεύνησης, προσπαθούμε να επιτύχουμε την πιο σύγχρονη δυνατή συμφωνία με τη Χιλή σε όλους τους τομείς. Αυτό περιλαμβάνει και τη βιώσιμη ανάπτυξη και το πολύ νέο ζήτημα η εμπορική ατζέντα. Ελπίζουμε ότι θα επιτύχουμε υψηλές φιλοδοξίες, ε, διότι όπως ε, είπε μόλις ο πρέσβης, ε, είναι έτοιμοι να επιτύχουμε μια συμφωνία που θα βρίσκεται, θα είναι καινοτόμο σε θέματα εμπορικής πολιτικής. Η διαφάνεια, πολύ σημαντική. Επίσης εκεί ακολουθούμε τις πιο σύγχρονες και πρόσφατες πρακτικές, θα δημοσιεύσουμε, θα δημοσιεύσουμε εκθέσεις, τις αρχικές διαπραγματευτικές μας προτάσεις και προσβλέπουμε να συζητήσουμε και με την ε, κοινωνία των πολιτών ε, και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, και ελπίζουμε να έχουμε ένα ψήφισμα το οποίο θα μας δώσει κάποια καθοδήγηση για το τι είναι σημαντικό για σας. Προβλέπουμε τη διοργάνωση εκδηλώσεων με την κοινωνία των πολιτών και μόλις ξεκινήσαμε Επαφή στη Χιλή μεταξύ της αντιπροσωπείας ε, και οργανώσεων ε, της Χιλής ώστε να έρθουμε σε επαφή με την κοινωνία των πολιτών στη Χιλή. Επίσης προσπαθούμε να δημοσιεύσουμε ε, τα έγγραφα, να δημοσιεύουμε τα έγγραφα στα ισπανικά. Μια σύντομη απάντηση στο ποια είναι η σύνδεση μεταξύ τη συμφωνία για τα βιολογικά προϊόντα και τη εξυγχρονισμένη συμφωνία. Κατά την άποψή μα, η συμφωνία αυτή είναι πολύ θετική. Είναι συμπληρωματική Δεν έχουμε πρόθεση αυτή η συμφωνία να περιλαμβάνει κάθε επιμέρους συμφωνία που έχουμε με την Χιλή. Οπότε και σε αυτή την περίπτωση έχουμε απλά μια συμπληρωματική συμφωνία. Τέλος, κάποια σχόλια σε σχέση με την βιώσιμη ανάπτυξη, με την ευρύτερη έννοια για τους ε, ε αυτόχθονες ε, είναι μία συμφωνία σύνδεσης ε, που σημαίνει ότι θα ασχολείται με πάρα πολλά ζητήματα. Ευχαριστώ πολύ. Και η συνάδελφος από την Γενική Διεύθυνση Γεωργίας θέλει να ε, σχολιάσει. Γεια σας, καλησπέρα σε όλους. Το όνομά μου είναι Ελένα Πανικίν. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες ο συζητήτρια κυρία Ροντρίγκε Πινιέρο έδωσε μια πολύ καλή επισκόπηση της συμφωνίας ε, για τα βιολογικά προϊόντα και απλά θα απαντήσω σε κάποιες ερωτήσεις για να κάνω κάποιε διευκρινήσει. Η πρώτη ερώτηση αφορούσε τη σύνθεση της Μικτής Επιτροπής Όπως αναφέρεται στο άρθρο 8 της συμφωνίας, η Μικτή Επιτροπή θα αποτελείται από ε, διόντως διορισμένους εκπροσώπους της ε, Ένωσης καθήκον της ε, θα είναι η διαχείριση της συμφωνίας, να λαμβάνει απόφαση υλοποίησης, να εξετάζει οποιοδήποτε αίτημα ή επικαιροποίηση για επέκταση νέα προϊόντα ή για ενισχυμένη συνεργασία. Η σύναψη της συμφωνίας προβλέπει ότι εκπρόσωποι της Κομισιόν θα λαμβάνουν εξουσιοδότηση να εκπροσωπούν την Ένωση στην Επιτροπή. Προβλέπεται ένας μηχανισμός για, την απλ για έναν εκπρόσωπο απλής ενημέρωσης των κρατών μελών στην Επιτροπή Βιολογικής Παραγωγής που θα λαμβάνει χώρα πέντε φορές, θα συναντάται πέντε φορές το χρόνο ε, και στο Συμβούλιο με πιθανή ένσταση ε, μιας ε, ε, που θα θέτει βέτο από τα κράτη-μέλη. Ένα άλλο ερώτημα ε, τι θα γίνει μετά από τρία χρόνια. Η συμφωνία προβλέπεται τώρα να τεθεί σε ισχύ και εφόσον δεν υπάρξει ένσταση από, τα, από οποιαδήποτε από τις δύο πλευρές θα παραταθεί ε, επα, επαόριστον εκτός αν το ένα μέρος ε, ενημερώσει το άλλο μέρος ότι ε, δεν επιθυμεί να συνεχιστεί. Δεν πρόκειται να γίνει εκτίμηση δικτύπου γι' αυτό. Απλά θα δούμε κατά πόσο προκύπτει οποιοδήποτε ζήτημα κατά τη διάρκεια αυτής της τριετίας. Μετά άκουσα κάποιες ανησυχίες σε σχέση με την ισοδυναμία και τη συμμόρφωση. Και στο πλαίσιο των σημερινών συζητήσεων στους τριμερείς διαλόγους για τον κανονισμό για τα βιολογικά. Εδώ θεωρώ ότι χρειάζεται να εξηγήσουμε λίγο τα ζητήματα αυτά. Μέχρι στιγμή το σύστημα λειτουργεί με δύο, είδους, ε, δύο ειδών εισαγωγέ. Αφενός ε, έχουμε ε, τρίτες χώρες με ισοδυναμία, δηλαδή τρίτες χώρες που έχουν ήδη αναγνωριστεί στο παρελθόν ως ισοδύναμες και μετά έχουμε ένα σύστημα ισοδύναμων ε, οργανισμών ελέγχου που ακολουθούν πρότυπα τα οποία έχουν αναγνωριστεί ως ισοδύναμα για την εισαγωγή βιολογικών προϊόντων. Τι θα αλλάξει με τη μεταρρύθμιση στο εξή. Οι οργανισμοί ελέγχου θα πρέπει να εφαρμοζούν τα ίδια πρότυπα Μπορούν να πιστοποιούν δηλαδή ως βιολογικά μόνο τα προϊόντα εκείνα που προέρχονται από παραγωγούς που έχουν εφαρμόσει τους βιολογικού κανόνες που εφαρμόζονται στην Ευρώπη. Αυτή είναι η έννοια τη συμμόρφωση. Από την άλλη πλευρά, φυσικά, εξακολουθεί να υπάρχει ισοδυναμία και στην εμπορική συμφωνία, αλλά μέχρι στιγμής οι ισοδυναμίε ε, υπήρχαν ε, μέχρι το 1992 και αυτού του είδους οι ε, συμφωνίες ε, εμπορίου ε, είναι νέες υπό την έννοια ότι δημιουργούνται για να ενισχύσουν την νομική βεβαιότητα αυτές τις τη ισοδυναμίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα μπορούν να κάνουν ο καθένας ό,τι θέλει. Φυσικά και όχι, διότι τα πρότυπα αξιολογούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από την αρμόδια αρχή της τρίτης χώρας, λαμβάνοντας υπόψη το ποια είναι αυτή η αρχή στη σε αυτή την περίπτωση. Θα αναλύει τον κατάλογο των προϊόντων, του κανόνε παραγωγή και θα ε, ε, πιστοποιεί την ισοδυναμία. Μια τελευταία πληροφορία σε περίπτωση που κάποια προϊόντα δεν θεωρούνται ισοδύναμα θα διαγραφούν από τη λίστα. Να κλείσω διότι μίλησα παραπάνω από το χώρο μου όσον αφορά τους ελέγχους του ΦΑΟ Φυσικά το ΦΑΟ θα ελέγχει, ελέγχει κάθε χρόνο τις ισοδύναμες τρίτες χώρες και φυσικά εφαρμοσμέτρα σε περίπτωση που ε, εντοπιστούν παρατυπίες. Για παράδειγμα, σε ορισμένε περιπτώσεις έχουν εξαιρεθεί ορισμένε κατηγορίες προϊόντων από την ισοδυναμία ή έχουν εφαρμοστεί διορθωτικά μέτρα μετά από αίτημα προς τις αρμόδιες αρχές για την πρόληψη περαιτέρω παρατυπιών. Ευχαριστώ. Μια σύντομη ερώτηση. Αν κατάλαβα καλά, δεν σχεδιάζεται να γίνει ε, μελέτη αντικτύπου. Γιατί? Πραγματοποιήθηκε μελέτη αντικτύπου στο παρελθόν. Στο πλαίσιο της ε, αναθεώρησης ε, του Γενικού Συστήματος Εμπορίου. Σχεδιάζουμε μετά από τρία χρόνια εφαρμογής τη εμπορική συμφωνία ε, να έχουμε μελέτη αντικτύπου, διότι δεν θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να γίνει μελέτη αντικτύπου εάν δεν διαπιστωθούν ελλείψεις ή επίμαχα θέματα. Εάν λοιπόν οι δύο πλευρές δεν θίξουν κάποιο συγκεκριμένο θέμα, η εμπορική συμφωνία θα συνεχίσει να ισχύει. Ευχαριστώ πολύ. Ίνμα, θέλεις να κλείσεις τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ όλους τους σκιώδεις συζητητές για αυτά που είπαν. Εννοείται και τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον πρέσβη φυσικά της Χιλής. Πιστεύω ότι όλοι συμφωνούμε για το ότι είναι μεγάλη η σημασία που έχει η ενίσχυση των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Χιλή, η οποία μοιάζει πολύ η Χιλή με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη από το 2003 λοιπόν προχωρούμε στην φιλοδοξία αυτή που θέλουμε να πετύχουμε. Τώρα χρειαζόμαστε ακόμα περισσότερο από ποτέ να εξυγχρονίσουμε την συμφωνία για να αντιμετωπίσουμε όλες τις σημερινές προκλήσεις. Καλά ρυθμισμένο εμπόριο, με κατάλληλο κεφάλαιο για την βιώσιμη ανάπτυξη, με τα στοιχεία τα οποία χρειαζόμαστε για να βοηθήσουμε την οικονομία της Χιλής ακόμα περισσότερο προς μια βιώσιμη ανάπτυξη, είμαι σίγουρη ότι θα κάνουμε ένα βήμα προς τα μπρος στη φιλοδοξία μας αυτή για να συγκεκριμενοποιήσουμε αυτή την εμπορική συμφωνία. Πιστεύω ότι και για τις δύο πλευρές είναι πολύ σημαντική η εμπιστοσύνη μεταξύ μας. Και εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα φροντίσουμε να υλοποιηθούν όλα όσα θέλουμε να συμπεριλαμβάνονται στη συμφωνία αυτή. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Η έκθεση θα είναι έτοιμη στις 19 Ιουνίου και θα έχουμε τη δυνατότητα τότε να συζητήσουμε, ενδεχομένω να υποβάλουμε τροπολογίες και στις 10 Ιουλίου κατά πάσα πιθανότητα θα ψηφίσουμε. Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ και περάμε στο σημείο 18 της μέρης της διάταξης, η εφαρμογή των διατάξεων της συνθήκης όσον αφορά τα εθνικά κοινοβούλια. Η ΑΦΚΟ είναι η αρμόδια επιτροπή. Θα θυμόσαστε ότι έχουμε ήδη συζητήσει για αυτό το θέμα όταν συζητήσαμε για τη ΣΥΤΑ, τη διαδικασία τροποποίησης. Και βέβαια στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την απόφαση της Σιγκαπούρης επίσης υπάρχουν κάποιες παρατηρήσεις σχετικά με το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων. Η συγκεκριτή μας είναι ο κύριος Όμπερμαγερ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κατά την χθεσινή διακυβερνητική κοινοβουλευτική συνάντηση συζητήθηκαν διάφορα θέματα τα οποία ε, σχετίζονται με την γνωμοδότησή μας. Θα ήθελα ε, να σημειώσω αυτά που συζητήθηκαν για τις εμπορικές συμφωνίες. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι ότι τα εθνικά κοινοβούλια δεν θα πρέπει να ε, είναι ένα βάρος, θα πρέπει να είναι ε, ένα όργανο με δημοκρατική νομιμοποίηση και θα πρέπει να γίνονται οι εργασίες ε, σύμφωνα με την ε, αξία και τη θέση των Εθνικών Κοινοβουλίων. κατά την ε, συζήτηση για τις διαπραγματεύσεις για τη Συμφωνία ΣΥΤΑ και την TTIP. Οι συμφωνίες αυτές διαπιστώνουμε ότι δεν είναι καθαρές εμπορικές συμφωνίες. και δεν ε, περιορίζονται στα κλασικά εμπόδια για το εμπόριο. Διαπιστώσαμε λοιπόν ότι υπάρχει ακριβώς ε, αυτός ο κίνδυνος σύγκρουσης ε, και το πρόβλημα ιεραρχίας εντός ε, των κρατών μελών. Στη δική μου πατρίδα την Αυστρία είδαμε κάτι τέτοιο, το είδαμε και στην Βαλονία. Επίσης ε, συζητήθηκε το EU Only ή η μεικτή ε, συμφωνία. Υπάρχουν ε, λοιπόν τα θέματα αυτά που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες που επικαλύπτονται και μπορέσαμε να συζητήσουμε και θέματα ορισμού. Η σχετική συζήτηση έχει γίνει και στο δημόσιο χώρο και σημειώνουμε ότι με τις συζητήσεις αυτές αμφισβητήθηκαν ε, και κάποιες βασικές αρμοδιότητες. Θέματα όπως είναι αυτό των ε, επενδύσεων και των ε, σχετικών δικαστικών μηχανισμών οδήγησαν ε, σε τέτοιες ε, συζητήσεις και καταλήγουμε στα εξή ε, συμπεράσματα ότι θέματα ορισμού στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα πρέπει να θίγουν τις αρμοδιότητες των κρατών μελών. Επίσης δεν θα πρέπει να αμφισβητείται η εκτελεστική εξουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε άλλωστε και την ε, συμφωνία της Σιγκαπούρης. Θα πρέπει εδώ να εξετάσουμε το θέμα της ευθύνης, διότι και εδώ οι αρμοδιότητες δεν είναι σαφώς διαχωρισμένες. Και γνωρίζουμε Άλλωστε, ότι στο πλαίσιο της συζήτησης για τα άρθρα 207 και 208 ε, από την Επίτροπο ε, ομολογήθηκε ότι υπάρχουν ε, ζητήματα διαχωρισμού, για να το πω με ήπια διατύπωση κιόλας. Υπάρχει εδώ σε μεγάλων συγκρούσεων σχετικά με το αν η ΣΥΤΑ είναι καθαρά Ευρωπαϊκή Συμφωνία ή εάν αποτελεί αρμοδιότητα και των κρατών μελών. Επίσης θα ήθελα να κάνω και κάποιες άλλες παρατηρήσεις. Η υποχρέωση συμμετοχής των κρατών μελών Ε, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στην ε, δημοκρατική διαδικασία. και τα κράτη-μέλη θα πρέπει επίσης να ενημερώνονται εξίσου με τους συναδέλφους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης, οι πολίτες είναι οι φορείς της δημοκρατίας, γι' αυτό θα πρέπει η διαφάνεια να ισχύει και για αυτούς. Αυτή λοιπόν είναι μια έκκληση που αξίζει να συζητηθεί. Οι συζητήσεις ε, θα πρέπει να οδηγούν σε ε, ψηφοφορία, σε δέσμες κιόλας, διότι είναι θέματα αυτά τα οποία συχνά οδηγούν σε περιπλοκές. Επίσης, πιστεύω ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εξετάσουν τις δικές τους εσωτερικές συνταγματικές δομές. Ε, είδαμε τι συνέβη στο Βέλγιο. Και νομίζω ότι έχω καταλάβει σωστά ότι η συνεργασία σε θέματα προστασίας καταναλωτών και σε περιβαλλοντικά θέματα. Μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ομάδες εργασίας όπου να συμμετέχουν ε, τα διάφορα κρατημέλη και τα κοινοβούλια τους. Αυτά όσον αφορά τις πρώτες προτάσεις για γνωμοδότηση της Επιτροπής μας. Προσβλέπω σε καλή συνεργασία. Και Προσβλέπω και στην καλή συνεργασία με του συναδέλφους από τι άλλε πολιτικές ομάδες και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Δίνω το λόγο στου σκιώδει εισηγητές, τον κύριο Βαλέζα από το ΕΛΚ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αντικαθιστώ τον Κρίστοφερ Φιέλνερ σήμερα. Εκ μέρου του θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την παρουσίαση αυτή. Όσον αφορά το θέμα αυτό, πρέπει να γνωρίζουμε σαφώς ότι είμαστε μια ένωση νόμων. Το ζήτημα των αρμοδιοτήτων της Ένωσης διέπεται από τις συνθήκες. Η εμπορική πολιτική είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έτσι έχουμε γίνει πιο ισχυροί και έχουμε μεγαλύτερη ευημερία. Σε δύο εβδομάδες ε, το δικαστήριο πρόκειται να ξεκαθαρίσει τα πράγματα για το που, ε, ποια είναι η διαχωριστική γραμμή των αρμοδιοτήτων όσον αφορά τις εμπορικές συμφωνίες και αναμένω είναι επιμερισμένες και οι αποκλειστικές αρμοδιότητες. Το κοινοβούλιο αυτό είναι το δημοκρατικά εκλεγμένο σώμα που αποφασίζει για τα θέματα αυτά. Όταν υπάρχει ε, επιμερισμένη ε, αρμοδιότητα όπως η ε, Συμφωνία τρικής Σχέσης με τις χώρες ACP, ο ρόλος του Κοινοβουλίου μας είναι μεγαλύτερος και πράγματι μπορεί να συμμετέχει. Εγώ ευχαρίστω να ακούσω προτάσεις για το πώς μπορεί να γίνει αυτό. Επίσης θεωρώ ότι δεν υπάρχει λόγος να βιαστούμε να τελειώσουμε αυτή την έκθεση, τη γνωμοδότηση δεδομένων των καθυστερήσεων στην Επιτροπή ΑΦΚΟ. Ε, ο Ο κύριο Σίλβα Περέρα, φυσικά είμαστε εδώ για να συζητήσουμε τις διατάξεις της συνθήκη όσον αφορά τα Εθνικό Κοινοβούλια ε, σε θέματα εμπορικά. Θέλω να υπενθυμίσω ότι με τη συνθήκη της Λισαβόνα ενισχύθηκε το εμπόριο ως ε, αποκλειστική αρμοδιότητα, περιλαμβάνοντας νέους τομείς όπως τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δεσμευτεί πλήρως για την χαράξη των νέων εμπορικών πολιτικών και έχει νόημα η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαπραγματεύεται μαζικά εμπορικές ε, συμφωνίες ε, επειδή είναι ισχυρότερη ε, από ότι τα επιμέρου κρατη κράτη-μέλη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που εκπροσωπεί τους πολιτέ τη Ευρωπαϊκής Ένωση στο πλαίσιο αυτό έχει να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο σε θέματα δημοκρατικής εξέτασης της εμπορικής πολιτικής και πιέζει για περισσότερη διαφάνεια και ενημέρωση του κοινού. Ε, έτσι δίνεται στην εμπορική πολιτική, ε, υπάρχει δημοκρατική νομιμότητα και ενισχύεται και η πτυχή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Στις εμπορικές συμφωνίες που αφορούν αποκλειστικά αρμοδιότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα Εθνικά Κοινοβούλια δεν συμμετέχουν άμεσα καθήκον τους είναι απλά να εξετάζουν ε, τη θέση της κυβέρνησής τους στο Συμβούλιο. Παρόλα αυτά, όταν οι συμφωνίες έχουν ευρύτερη κάλυψη και είναι ε, μικτές συμφωνίες, ε, καλύπτουν δηλαδή ζητήματα με αποκλειστικές αρμοδιότητες ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών μελών, είναι απόλυτο αιτιολογημένο ότι τα εθνικά κοινοβούλια θα συμμετέχουν πλήρως οι κυβερνήσει πρέπει να συζητούν και να διανέμουν τις πληροφορίες που έχουν λάβει από, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τι εμπορικέ διαπραγματεύσει και τι εμπορικέ συμφωνίε στα εθνικά τους κοινοβούλια. Τελικά, αυτού του είδου συμφωνίες θα ακολουθήσουν τη συνήθεια διαδικασία εκύρωσης. Όπως γνωρίζετε η επερχόμενη απόφαση του δικαστηρίου περί θέματων αρμοδιότητας εκύρωσης της ε, εμπορικής συμφωνίας με τη Σιγκαπούρη θα ξεκαθαρίσει ελπίζουμε τη φύση των εμπορικών συμφωνιών. Έχουμε τη γνωμοδότηση για την συμφωνία ε, της Σιγκαπούρης ε, του Γενικού Εισαγγελέα από το 2016, αλλά αναμένουμε την τελική απόφαση του δικαστηρίου. Αφού θα έχουμε αυτή την απόφαση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να σκεφτούν ποιο θα είναι το μελλοντικό ε, αντικείμενο των ευρωπαϊκών εμπορικών ε, συμφωνιών. Το σημαντικότερο κατά την άποψή μου είναι να διασφαλίσουμε την ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, να δρά στο εμπορικό επίπεδο, να έχει μια εμπορική ατζέντα νομιμοποιημένη δημοκρατικά, βασισμένη σε αξίες και τέλος μια εμπορική ατζέντα που θα οδηγήσει σε καλά αποτελέσματα και ευκαιρίες. Τέλος, πέραν όλων αυτών, αυτή η εμπορική ατζέντα, αυτό το εμπορικό θεματολόγιο θα πρέπει να εξελίσσεται διαρκώς, να γίνεται όλο και πιο διαφανές και φυσικά εκεί τα εθνικά κοινοβούλια και οι πολίτες ε, θα υποφεληθούν από τα νέα επίπεδα διαφάνειας στις εμπορικές διαπραγματεύσεις που πρέπει να συνεχίσουμε να ε, βελτιώνουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Τάρμ δεν είναι εδώ. Η κυρία Σάκε δεν είναι εδώ. Ο κύριος Σόλτς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να σημειώσω ότι τα κράτη-μέλη στο πλαίσιο της ε, συνθήκης ε, της Λισαβόνας ε, έχουν χωρίσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση την αρμοδιότητα για τα εμπορικά θέματα. Θα πρέπει λοιπόν να ελέγχουν και να παρακολουθούν αυτόν τον πυλώνα της ευρωπαϊκής πολιτικής. Και να ενεργούν αντίστοιχα στις περιπτώσεις των οριζοντίων συμφωνιών. Και εμείς κατά τη λήψη των αποφάσεών μας ε, θα πρέπει ε, να φροντίζουμε για τη συμμετοχή των κρατών μελών. Είναι θέμα ευθύνης και ενίσχυσης της δημοκρατικής συμμετοχής. Θα ήθελα να κάνω και μια δεύτερη παρατήρηση. Χθες Ακούστηκε αυτό στην ε, ακρόαση της ε, ΙΜΚΟ. Που, της ΑΦΚΟ. Πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Ε, καθηγητής από το Πανεπιστήμιο Χούμπολτ είπε πολύ σαφώς ότι τα ερωτήματα που τίθενται αυτή τη στιγμή στα κράτη-μέλη τη συζήτηση αυτή θα πρέπει να την εκμεταλλευτούμε και στον διάλογο με τα εθνικά κοινοβούλια και άλλους φορείς, αλλά και με την κοινωνία και τους φέρονται στην ευθύνη. Η έκθεση αυτή είναι ιδιαίτερα επίκαιρη. Περιμένουμε την απόφαση του δικαστηρίου για την Συμφωνία της Σιγκαπούρης. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε τον επιμερισμό των αρμοδιοτήτων. Περιμένουμε λοιπόν την απόφαση να δούμε πώς θα προχωρήσουμε από εδώ και μπρος. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πεκίν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Το θέμα των Εθνικών Κοινοβουλίων είναι ευρύτερο από ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Προκείται για την ίδια την ουσία της δημοκρατίας στην Ευρώπη δημοκρατία που είναι πλήρη, συνάδελφοι, μόνο όταν υπάρχει επιμερισμός των εξουσιών σε κάθε επίπεδο ε, ε, κυβερνητικό που αντιστοιχεί σε διαφορετικό έλεγχο του λαού, ε, ένα κοινοβούλιο αντιστοιχεί σε ένα λαό, ένα δημοτικό συμβούλιο, σε ένα δήμα. Αλλά όταν αποφασίζει κανείς να μεταφέρει στις Βρυξέλλες την αρμοδιότητα διαπραγμάτευση εμπορικών συμφωνιών, δίνει την εξουσία αυτή σε μια μη αιρετή κυβέρνηση ε, και ακόμη και αν υπάρχει ενίσχυση των ελέγχων, ναι, εντάξει, έχουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά δεν αντιστοιχούν, αυτά δεν συγκρίνονται με τα όσα συμβαίνουν σε ένα ε, εθνικό κοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά από τη Λισαβόνα είναι πιο ισχυρό, αλλά όσον αφορά τι συμφωνίε ελευθέρων συναλλαγών, ε, θα έπρεπε να λαμβάνει την υποστήριξη των εθνικών κοινοβουλίων για να γίνονται σεβαστέ οι επιθυμίε των πολιτών. Πολλέ φορέ έχει αποδείξει η Κομισιόν ότι δεν λαμβάνει υπόψη άποψη, την άποψη του Ευρωκοινοβουλίου όπως σε θέματα ε, συμφωνιών όπως έγινε με τις συστάσεις μας για το ΤΕΖΑ. Για παράδειγμα, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν συνάδουν οι πράξεις του με τις συνθήκες. Το άρθρο 107, στο οποίο βασίζεται η εμπορική πολιτική της Ένωσης, αναφέρεται σαφώς ε, η θέση του Κοινοβουλίου. Οι συνθήκες προβλέπουν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θα πρέπει να διαβουλεύεται διαρκώς στο Συμβούλιο, αλλά Θεσπίζουν επίση ότι οι υποχρεώσει τη Κομισιόν προ το Ευρωκοινοβούλιο συνίστανται σε μια απλή αναφορά και εμεί οι συνάδελφοι γνωρίζουμε ε, τι είναι αυτέ οι αναφορέ. Χρειάζεται λοιπόν ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στι συνθήκε αλλά σε κάθε περίπτωση ο ρόλος των ε, εθνικών κοινοβουλίων δεν πάβει να είναι απαραίτητος για να υπάρχει ένα επιπλέον επίπεδο δημοκρατικού ελέγχου πάνω από την Κομισιόν, κυρίως στις τελικές φάσεις, δηλαδή αφού το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο έχουν εκφέρει την άποψή τους. Θεωρώ, συναδέλφοι, ότι πρέπει να καταλήξουμε σε, σε καλύτερο ορισμό των μεικτών ε, ε, συμφωνιών όπου να μην μπορεί η Κομισιόν να έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης και το Συμβούλιο να κάνει κάτι άλλο. Αυτό είναι απαραίτητο για να φυλάξουμε τα προνόμια των κρατών μας αλλά και για να διατηρήσουμε μια κυριαρχία και έναν έλεγχο, διότι αλλιώς θα λαμβάνονται οι αποφάσεις στα ψηλά επίπεδα, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι πολίτε, οι οποίοι αισθάνονται όλο και περισσότερο το δημοκρατικό έλλειμμα στην Ευρώπη. Ε, άκουσα με ενδιαφέρον τις απόψεις του εισηγητή και ελπίζω να συμμετέχω και εγώ και να συμβάλλω σε αυτό το θέμα που θεωρώ πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστώ. Κύριε Καρίμ, θέλετε το λόγο, όχι. Παρακαλώ, κύριος Μάρτιν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν ήθελα να πάρω το λόγο. Ε, αλλά άκουσα την τελευταία παρέμβαση της κυρίας Πεκίν και νομίζω ότι κάνει λάθος. Εάν όλοι ε, έχουν την ευθύνη, κανείς δεν έχει την ευθύνη και με 30 και κοινοβούλια, θα ε, καταλήξουμε σε αδιέξοδο. Νομίζω λοιπόν ότι η συνθήκη της Λισαβόνας εδώ είναι σωστή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει την εντολή από τα κράτη-μέλη, από τις ε, εκλεγμένες κυβερνήσεις και τα εθνικά κοινοβούλια θα πρέπει τότε σε αυτό το στάδιο να ελέγξουν την εντολή. Με την έναρξη των διαπραγματεύσεων τον ρόλο αυτό θα πρέπει να αναλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης, θα πρέπει να υποβάλλονται εκθέσεις μετά από κάθε γύρο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σε αντίθεση με, αυτά που μόλις ακούσαμε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν συμφωνεί με όλα όσα λέμε, δεν κάνει όλα όσα λέμε, αλλά ακούει τη θέση μας ε, και στο τέλος της διαδικασίας αυτής, αν δεν μας έχουν ακούσει αρκετά προσεκτικά, ε, έχουμε το δικαίωμα να απορρίψουμε το αποτέλεσμα και το ξέρει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν λέω ότι θα πρέπει να συμπίπτουν οι δύο αυτές θέσεις, ε, διότι δεν λειτουργεί έτσι η δημοκρατία, αλλά θα πρέπει να γνωρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι αν ξεφύγει πολύ από την εντολή μας, τότε θα απορρίψουμε τη θέση της και τα ε, ε, εθνικά κοινοβούλια θα πρέπει να ε, εγκρίνουν την εντολή και φυσικά υπάρχει χώρος για τακτικές επαφές, για ενημέρωση των κοινοβούλιων. Αλλά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τελικά θα πρέπει να δίνει την έγκριση όχι. Σύντομη παρέμβαση του κυρίου Σόλτς. Μία μικρή ερώτηση ή ε, μια μικρή ανταλλαγή απόψεων θα ήθελα με τον Ντέιβιτ, διότι συμφωνώ με αυτό που μόλις ε, είπε. Αλλά το να δώσουμε το δικαίωμα πρωτοβουλίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα μας έδινε την ευκαιρία να εισάγουμε διαφορετικό περιεχόμενο στην διεθνή εμπορική πολιτική και έτσι να ενισχύσουμε και τη δημοκρατική συμμετοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων. Επιτρέψτε μου να, απαντήσετε, να, να απαντήσω. Ναι, εμένα θα μ' άρεσε κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι σημαντικό ε, κενό στην ε, συνθήκη της Λισαβόνα είναι ότι δεν έχουμε εμείς επίσημο ρόλο στην διαπραγμάτευση της εντολής ε, και συμφωνώ ότι κάτι τέτοιο θα ήταν ένα σημαντικό βήμα πρόοδου. Ωραία. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διαφορετική άποψη. Μήπως θα ήθελε να μας ε, την αναπτύξει. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Είμαι από την διοργανική, από το διοργανικό τμήμα της Digitrade. Κάποια από αυτά που είχα εγώ να σας πω, τα είπαν οι ευρωβουλευτές ακόμα καλύτερα από ό,τι θα τα έλεγα. Πάντως, είμαστε στα μέσα του δρόμου για την εντολή της Επιτροπής. Έχουμε αναλάβει δέσμευση για συνεργασία με τα Εθνικά Κοινοβούλια και για πιο αποτελεσματική και εντατική συνεργασία μεταξύ μας. Αυτό διευκρινίζεται ήδη από το 2015 στην ανακοίνωσή μας «Εμπόριο για όλους» που έχουμε ήδη συζητήσει. Επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υπογραμμίσει ότι θα κάνει περισσότερες προσπάθειες προκειμένου να γίνεται συζήτηση για αυτές τις συμφωνίες στις χώρες μέλη και να υπάρχει διάλογος με τις κοινωνίες των πολιτών. Δεσμεύτηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης να πηγαίνει τακτικά στις χώρες μέλη και στα εθνικά κοινοβούλια για να συζητά εμπορικά ζητήματα. Και οι εθνικές κυβερνήσεις ζητούμε να είναι πιο δραστήριε στις συζητήσεις που γίνονται για το εμπόριο. Κατόπιν όλων αυτών δημοσιεύσαμε υλικό στο διαδίκτυο για εμπορικέ συμφωνίε, για παράδειγμα εκθέσεις για διάφορους διαπραγματευτικούς γύρους, για προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, νομικά κείμενα προς συμφωνία, κάτι το οποίο έχει επιτρέψει καλύτερη ενημέρωση. Και όλα αυτά πέρα βέβαια από τις υποχρεώσεις που έχουμε έτσι και αλλιώς αναλάβει, που είναι να ενημερώνουμε πλήρως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις διαπραγματεύσεις μας. Συνεπώς υπάρχει ενημέρωση και προς το κοινό και προς τους εκπροσώπους των χωρών μελών, ε, Συμβούλιο, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πιστεύουμε λοιπόν ότι κατόπιν όλων αυτών θα μπορέσουμε να έχουμε καλύτερες σχέσεις ακόμα και με το κοινό, την κοινωνία των πολιτών, αλλά και με τα εθνικά κοινοβούλια όσον αφορά εμπορικές συμφωνίες. Τώρα μπορούμε βέβαια να βάλουμε σε κατηγορίες τις εμπορικές συμφωνίες, είτε επιμερισμένης αρμοδιότητας είτε αποκλειστικής. Δεν είναι το ίδιο αυτές οι δύο κατηγορίες, δεν ελέγχονται με τον ίδιο τρόπο δημοκρατικά οι συμφωνίες αυτές. Αυτό είναι κάτι το οποίο υπόθηκε ήδη. Τώρα όσον αφορά τις συναντήσεις που είχε επίτροπος με τα Εθνικά Κοινοβούλια για να συζητήσει την εμπορική πολιτική είναι κάτι το οποίο εκτιμήθηκε όλος ιδιαίτερος. Πρέπει να δούμε βέβαια τα συμπεράσματα από την γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Θα πάρει χρόνο να αναλύσουμε τις επιπτώσεις αυτής της απόφασης, της γνωμοδότησης μάλλον. Αλλά έτσι θα διευκρινιστούν πολλά ζητήματα, κάτι που είναι θετικό για όλους μας, όλους εμάς που ασχολούμαστε με την εμπορική πολιτική. Ευχαριστούμε ο κύριος Όμπερμαϊρ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σύντομα, ευχαριστώ για τις επικοδομητικές παρεμβάσεις. Θα δούμε πώς μπορούμε να τα συμπεριλάβουμε αυτά στην πράξη. Πάντως, ε, γεγονός παραμένει ότι υπάρχει ανάγκη για συζήτηση. Επίσης, τονίστηκε ότι είναι σημαντική η επαφή με τα εθνικά κοινοβούλια. Και από την διαδικασία για την Συμφωνία ΣΕΤΑ μάθαμε πολλά και μπορούμε να μάθουμε ακόμα πολλά. Ε, συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι θα πρέπει να ενεργήσουμε με βάση τη συνθήκη της Λισαβόνας. Είναι σημαντικό να υπάρχουν επαφές και νομίζω ότι έχουμε αρκετό υλικό για να ξεκινήσουμε την εργασία πάνω στο θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Στις 19-20 Ιουνίου θα συζητήσουμε την έκθεσή σας. Και θα, πρέ... θα ενδεχομένως και, και τροπολογίες. Έτσι φτάνουμε στο σημείο 19 και να σας θυμίσω ότι έχουμε και το σημείο 20 που είναι σημαντικό θέμα προς συζήτηση στην ε, ημερησία διάταξή μας. Να προχωρήσουμε λοιπόν γρήγορα. Το σημείο 19 είναι προφορική ερώτηση και ψήφισμα για την εφαρμογή του Συμφώνου Βιωσιμότητας στον Μπαγκλαντές. Επανειλημμένα το έχουμε συζητήσει αυτό και στο πλαίσιο του ψηφίσματος ε, για τα υφάσματα. η ασφάλεια των κτηρίων, η πυρασφάλεια στο Μπαγκλατές, βελτίωση της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτά είναι θέματα που μας ενδιαφέρουν. Και λαμβάνουμε πληροφορίες ότι στο πλαίσιο του συμφώνου έχουμε στενή συνεργασία ανάμεσα σε αρχές αλλά και άλλους φορείς. Για παράδειγμα, στο θέμα του ελάχιστου μισθού, αλλά και το δικαίωμα συλλογικών διαπραγματεύσεων ε, των εργαζομένων σε περιπτώσεις απολύσεων. Απομένει λοιπόν αρκετή δουλειά στο θέμα αυτό. Η Κομισιόν τον Μάρτιο ε, ζήτησε τήρηση του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων και τόνισε το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η επόμενη συνάντηση των εταίρων του Συμφώνου θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο και το Διεθνές Γραφείο Εργασίας ε, θα οργανώσει την ε, ετήσια ε, διάσκεψή του με ειδική ε, συζήτηση για το Μπαγκλαντές. Προφορική ερώτηση λοιπόν και ψήφισμα και δίνω το λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο Κάριν, παρακαλώ. Um, Ευχαριστώ πολύ. Το Μπαγκλαντές έχει αλλάξει πάρα πολύ τα τελευταία 30 χρόνια και μπορούμε να είμαστε περήφανοι για το ότι η ευρωπαϊκή εμπορική πολιτική αποτέλεσε ένα σημαντικό παράγοντα για την αλλαγή αυτή. Ακόμα βέβαια και αν 6 εκατομμύρια άνθρωποι παραμένουν πάρα πολύ φτωχοί, η αλλαγή είναι τεράστια είναι δεύτερη μετά την Κίνα στις εξαγωγές. Το Μπαγκλαντές έχει προχωρήσει πάρα πολύ τα τελευταία 10 χρόνια. 28,1% δισεκατομμύρια ήταν το πλεόνασμα που είχε, το που είχε τον Μπαγκλαντές, αλλά σε αυτό συμμετέχουν πάρα πολλοί γυναίκες οι οποίες αποτελούν το 70% του εργατικού δυναμικού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνεισφέρει λοιπόν. Η κλώστη φαντουργία συνεισφέρει πάρα πολύ με δασμού σε ολόκληρο τον κόσμο και η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε μονομερός να επιτρέψει πρόσβαση χωρίς δασμούς στην εσωτερική της αγορά προϊόντων, μεταξύ άλλων της κλωστιφαντουργία. Αυτή η προτιμησιακή γενναιόδορη μεταχείριση βοήθησε πάρα πολύ τις αλλαγές στον Μπαγκλαντές. Όμως η συμφωνία τώρα αυτή γενικών προτιμήσεων συν αποτελεί ένα βήμα παραπάνω γιατί βασιζόμαστε σε εμπόριο βάση αξιών και αρχών. Δηλαδή εμείς συζητούμε από τους εμπορικούς μας εταίρους να σέβονται βασικές αρχές στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των εργασιακών δικαιωμάτων. Όντως η ασφάλεια έχει ουσιαστικά βελτιωθεί, όμως παρόλα αυτά καταραίουν κτίρια και συμβαίνουν και άλλες καταστροφές στην κλωστιφαντουργία, στα εργοστάσια δηλαδή τα τελευταία χρόνια. Οπότε ήταν απόλυτα θεμητό οι Ευρωπαίοι καταναλωτές να ζητούν από τον Μπαγκλαντές να τηρεί όσα πρέπει να τηρεί για την ασφάλεια των εργαζομένων και τα δικαιώματά τους. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Διεθνή Οργάνωση Εργασίας και άλλους σημαντικούς εταίρους, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά, αλλά και με την κυβέρνηση του Μπαγκλαντές, κάθισε και συζήτησαν πώς θα βελτιωθεί η ασφάλεια και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Εξού και προέκυψαν αυτές οι θετικές αλλαγές. Πάνω από 200 ε, ξένες μάρκες έχουν υπογράψει διάφορες συμφωνίες ασφάλειας για την πυρασφάλεια, την ασφάλεια των ε, κτίριων, την ασφάλεια των εργαζομένων στον Παγκλαντές και υποσχέθηκαν να ξοδέψουν δεκάδες εκατομμύρια για να βελτιωθεί η ασφάλεια στους χώρους εργασίας. Εμείς πρέπει να στηρίξουμε τις ε, πρωτοβουλίες αυτές του ιδιωτικού τομέα και να ενθαρρύνουμε ακόμα περισσότερο τις επιχειρήσεις, γιατί είναι και προς το δικό τους συμφέρον, βελτιώνεται η εικόνα τους προς τα έξω. Και η ανταγωνιστικότητά τους επίσης ε, μέσα στην παγκόσμια κατάσταση. Όσον αφορά την ε, ασφάλεια των εργαζομένων πάντως, αυτό δεν είναι το μόνο ζήτημα που πρέπει να εξετάσουμε όταν συζητάμε την συμφωνία αυτή γενικών προτιμήσεων ε, ενισχύεται το εμπόριο εξαιτίας της ανταγωνιστικότητά του, εξαιτίας της οικονομίας κλίμακας. Πάντως παρά την αύξηση των πωλήσεων και την ανάπτυξη της οικονομίας των Μπαγκλαντές, 67 δολάρια είναι ο μέσος όρος μηνιαίου μισθού από το 2016. Υπάρχουν βέβαια και άλλες τάσεις τα τελευταία χρόνια. Από το Δεκέμβριο του 2016 απολύονται εργαζομένοι, συνδικαλιστές συλλαμβάνονται, διώκονται, φυλακίζονται και δεν γίνονται μεταρρυθμίσεις όσον αφορά τα εργασιακά δικαιώματα. Το κλίμα γενικά έχει επιδεινωθεί όσον αφορά τους εργαζόμενους και τα δικαιώματά τους. Συνεπώς, η κυβέρνηση του Παγκλαντές πρέπει να κάνει περισσότερα. Είναι ένα εσωτερικό ζήτημα για να υπάρξει ελευθερία του συνεταιρίζεσθε, η προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και των ε, εκπροσώπων τους τα συνδικάτα και η δημιουργία τους πρέπει να διευκολύνεται, να εφαρμόζονται καλύτερα οι νόμοι που ήδη υπάρχουν και να μην ε, διώκονται οι συνδικαλιστές, αλλά αντίθετα αυτοί που διώκονται τους συνδικαλιστές να τιμωρούνται. Έτσι λοιπόν θέλουμε να βοηθήσουμε την κυβέρνηση του Πακλαντές, τις ε, ιδιωτικές εταιρείες και την διεθνή κοινότητα. Και χαιρόμαστε και εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για τη συμφωνία ανάμεσα στον ιδιωτικό τομέα και το Μπαγκλαντές. Η επιχειρήση και η οικονομία του Μπαγκλαντές μπορεί να είναι επιτυχής εφόσον γίνουν περισσότερα πράγματα και εφαρμοστούν καλύτερα οι νόμοι. Τώρα έχουμε φτάσει σε ένα σταυροδρόμι. Οπότε, συνάδελφοι, που περνάμε το μήνυμα στην κυβέρνηση του Μπαγκλαντές και όλους τους αδιαφερόμενους ότι θέλουμε περισσότερες προσπάθειες για να υπάρξει πρόοδος όσον αφορά την, ε, το σύμφωνο βιωσιμότητας και να μην δεχτούμε παραβιάσεις των δικών μας ε, αρχών. Το 2018 το Μάιο εκπνέει η συμφωνία, αλλά προς το παρόν δεν έχουν επιτευχθεί όλοι οι στόχοι. Εμείς θέλουμε να πετύχει το Παγκλαντές και να συνεχίσει στο δρόμο της βιώσιμης ανάπτυξης και θέλουμε και τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Σύμφωνο Βιωσιμότητας να πετύχουν για να έχουμε εμπόριο που βασίζεται σε αξίες και αρχές. Και οι εταιρείε οι οποίες ε, δραστηριοποιούνται στο Μπαγκλαντές και που έγιναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τα τελευταία χρόνια και που προσφέρουν καλές τιμές και καλά προϊόντα στους καταναλωτές να δραστηριοποιούνται σύμφωνα με τις δικές μας αξίες και των καταναλωτών μας. Πρέπει να ενισχύσουμε λοιπόν τις προσπάθειές μας για να γίνει αυτό πραγματικότητα και γι' αυτό η Επιτροπή Διεθνούς Μπορεί αποφάσισε να προτείνει προφορική ερώτηση που συνοδεύεται από ψήφισμα για να αναφερθούμε στις σημερινές αδυναμίες. Προσβλέπω σε συνεργασία με όλους τους συναδέρφους, όπως πάντα, για το ψήφισμα αυτό και ευχαρίστως να συμπεριλάβω και όλα τα μέτρα τα οποία θα ήθελαν να αναφερθούν στο ψήφισμα αυτό οι συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Καρύμ. Πέντε λεπτά έχουμε για το θέμα αυτό. Σας παρακαλώ λοιπόν ένα λεπτό χρόνο ομιλίας ο καθένας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Καράν για τις προσπάθειες που έχει καταβάλει για το θέμα αυτό. Θα ήθελα να αναφέρω κάποια σημαντικά γεγονότα. Τέσσερα χρόνια έχουν περάσει από το τρομακτικό ε, ατύχημα στο Μπαγκλαντές ε, και εκτιμάται το 2016 εκατοντάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε εργοστάσια του Μπαγκλαντές 12.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε ατυχήματα και πάρα πολλοί άλλοι χάνουν τη ζωή τους λόγω ασθενειών ε, στον τόπο εργασία στο Μπαγκλαντές. Πρέπει να μας ανησυχήσει αυτό και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο για να μειωθούν οι θάνατοι αυτοί. αυτό γίνεται να επιτευχθεί με ένα θετικό τρόπο, με μια συμφωνία βιώσιμης παραγωγής ε, για να προστατευτούν οι εργαζόμενοι, ειδικότερα στον τομέα των έτοιμων ενδυμάτων. Στην τελευταία αξιολόγηση κατέστησε σαφές ότι έχουν γίνει βελτιώσεις κυρίως σε θέματα πυροπροστασίας. Επίσης εφαρμόστηκαν διορθωτικά μέτρα ε, για κρίσιμα ζητήματα ασφαλείας. Η μεγαλύτερη δυσκολία κατά την άποψή μας εξακολουθεί να είναι το ζήτημα των εργασιακών δικαιωμάτων ειδικότερα η αλλαγή της εργασιακής νομοθεσίας που έγινε από το 2013, η εφαρμογή των συμφωνιών της Διεθνούς, Διεθνούς Οργανούς Εργασίας και η σωστή κατάρτιση ενός καταλόγου συνδικάτων. Το μήνα αυτό επικτείνει μια συνάντηση στην ΤΑΚΑ που θα είναι κρίσιμη σημασία για να δούμε αν το Μπαγκλαντές θα συνεχίσει να συμμορφώνεται ε, με τη συμφωνία αυτή και τις λοιπές. Ε, δηλαδή κατά πόσο θα συνεχίσει να υποφελείται ε, από, τις, από το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων και από τη συμφωνία τα πάντα πλην όπλων. Αυτό που είναι σημαντικό κύριε Πρόεδρε στην περίπτωση του Μπαγκλαντές είναι να σημειωθεί κάποια πρόοδος. Έχουμε ένα εξαιρετικό ψήφισμα εδώ το οποίο εκφράζει τις κύριες ανησυχίες μας, τις κύριες δυσκολίες και παραθέτει τα βασικότερα ζητήματα που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ώστε να βεβαιωθούμε ότι υπάρχει συμμόρφωση με το σύμφωνο βιωσιμότητας ε, έως ότου εκπνεύσει. Και φυσικά η παράταση είναι βεβαιό κατά πόσο θα χορηγηθεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εκ μέρους του Άγγλου Γραμμύρας ε, θα σας μιλήσω, θα μιλήσω λίγο πιο γρήγορα, ε, πιο πολύ από ότι προβλεπόταν. Ήθελε αρχικά να ευχαριστήσει τον κύριο Καρύμ για τις προσπάθειές του και ευχαριστεί που έλαβε υπόψη πολλές από τις συστάσεις της, αλλά την προβληματίζει το ότι δεν ε, ε, ε, συνεργαστήκαμε άμεσα για τη σύνταξη της, ε, του ψηφίσματος, αλλά είναι ικανοποιημένη από αυτό. Γενικά υποστηρίζει το ψήφισμα, θεωρεί ότι είναι εξαιρετικό ότι επισημαίνει τον τομέα των έτοιμων ενδιαμάτων και πόσο σημαντικό είναι ο τομέα για την ανάπτυξη των Παγκλαντέ και φυσικά την προσοχή στα πολλά σοβαρά προβλήματα του τομέα. Ωστόσο, θεωρεί ότι δεν αναφέρεται το ζήτημα ως αρκετά επίγον αν το συγκρινούμε με την επιστολή που έστειλε Γενική Διευθυν... Ε, έστειλαν κάποιες γενικές διευθύνσεις στην κυβέρνηση του Μπαγκλαντές τον Μάρτιο ε, δεδομένων των όσων αναμένουμε να γίνουν στην διάσκεψη του ILO ε, πιστεύει ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη περισσότερο τις δηλώσεις της Κομισιόν στο ψήφισμα για πιθανές συνέπειες όσον αφορά τις πρόσβαση στην αγορά του Μπαγκλαντές και τις πρόσβαση του Μπαγκλαντές ε, στο σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων αν δεν αλλάξει διαδικασίες. Το ψήφισμα είναι καλό λοιπόν αλλά πιστεύει ότι πρέπει να είμαστε πιο σαφείς όσον αφορά τις επιπτώσεις που θα έχει στον Μπαγκλαντές ε, η μη πρόοδος προς καλύτερες συνθήκες. Ευχαριστώ κύριος. Κύριε Μινέρ. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Με εκπλήσω ο τόνος της έκθεσης είναι επικριτική αλλά όχι αρκετά. Όντως, βλέπουμε ότι το Μπαγκλαντές εξακολουθεί να μην τηρεί αυτά τα οποία πρέπει. Με τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις που λένε για τις παρεβιάσεις που γίνονται όσον αφορά τα ανθρώπινα και τα εργασιακά δικαιώματα, για τον μισθό των εργαζομένων που μειώνεται αντί να αυξάνεται. 61 ευρώ το μήνα παίρνουν κατά μέσο όρο μισθό οι κάτοικοι του Μπαγκλαντές. Δεν μπορεί να ζήσει κανείς με αυτά τα χρήματα, ούτε καν στον Μπαγκλαντές. Είναι ντροπή λοιπόν. Και εμείς φοράμε τα ρούχα που φτιάχνουν αυτοί οι άνθρωποι. Πολλοί κάνουν ε, απεργία, αλλά τους διώκουν στη συνέχεια, τους απολύουν τους ανθρώπους αυτούς. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να καθίσουμε και να σκεφτούμε. Το Μπαγκλαντές μπορεί να έχει πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά στα πλαίσια του όλα απόπλα με τέτοιες παραβιάσεις. Βέβαια, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τέλεια. Οι δικές μας επιχειρήσεις ζητάνε από τον Μπαγκλαντές να φτιάξουν τα ρούχα τους. Με αυτόν τον τρόπο δεν βελτιώνεται η κατάσταση στη χώρα. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα στην έκθεση να αναφέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα φροντίσει να τηρούνται οι κανόνες όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Μπαγκλαντέ. Αλλιώ να σταματήσουν αυτές οι σχέσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Σάντρα, σύντομα παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα σε όλους. Ας ξεκινήσουμε ευχαριστώντας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την υποστήριξή σας στο θέμα αυτό. Ελπίζουμε ότι θα μας βοηθήσει, διότι δεν είναι καθόλου εύκολο το θέμα αυτό. Είναι πολύ καλό το ότι έρχεστε σε επαφή με όλους τους ενδιαφερόμενους κύκλους και πρέπει να σας ε, ευχαριστήσω από το βάθη της καρδιάς μου για το θέμα αυτό. Επίσης, ε, κύριε Καρύμ, να σας ευχαριστήσω για το σχέδιο ψηφίσματος. Ε, πιστεύουμε ότι είναι ισορροπημένο με την έννοια ότι δείχνει τι θα πρέπει να κάνουν οι διάφοροι ενδιαφερόμενοι, ο ιδιωτικός τομέας, η διεθνής κοινότητα αλλά και η κυβέρνηση του Μπαγκλαντές που σίγουρα είναι σημαντικός παράγων στο θέμα αυτό. Θα ήθελα επίσης να πω ότι είναι ένα θέμα στο οποίο είναι ε, εξαιρετική και αποτελεί υπόδειγμα η συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ε, διότι ε, μιλάμε με μία φωνή και όπως υπόθηκε, θα πρέπει να στείλουμε ένα σαφές και ισχυρό μήνυμα, ώστε να καταλάβει η άλλη πλευρά τι περιμένουμε από αυτήν. Είναι λοιπόν σημαντικό για μας το ψήφισμα αυτό να είναι στοχευμένο και ε, να επικεντρώνεται στα βασικά. Είναι λοιπόν προτεραιότητα και δική σας και δική μας το θέμα αυτό. Θεωρούμε ότι το Μπαγκλαντές θα πρέπει να ασχοληθεί με τις συστάσεις που κρεμούν ακόμα. Γνωρίζουμε ότι η ελευθερία του συνεταιρίζεσθε είναι ιδιαίτερα επώδυνο θέμα, όπως και οι συλλογικές διαπραγματεύσεις. Θέλουμε και εμείς να θεωρήσουμε ότι η συνεργασία θα μπορέσει να συνεχιστεί και μετά από τη λήξη της προθεσμίας. Επίσης, Όσον αφορά την ε, υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, έχουμε συζήτηση με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας ε, και πιστεύουμε ότι η ενθάρρυνση του διαλόγου είναι ζωτική σημασίας, είναι επίσης ζωτική σημασίας να ασχοληθούμε με τις αγοραστικές πρακτικές. Δεν θέλω ε, να μακρηγορήσω, αλλά δεν είναι ένα θέμα το οποίο μπορούμε να ξεχάσουμε και να νύπτουμε τα σχήρας μας. Επίσης, ε, είναι θέματα τα οποία θίγουμε καθημερινά απέναντι στο ε, Μπαγκλατές, ε, όπως για παράδειγμα το θέμα της ελευθερίας του συνεταιρίζεστε. Θα ήθελα επίσης να πω ότι συμμερίζομαι απολύτως το συμπέρασμά σας για τις αξίες μας. Δεν μπορούμε να παρέχουμε προτιμησιακό καθεστώς χωρίς να είναι σαφές το τι περιμένουμε και δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να χορηγούμε τέτοιο καθεστώς εάν αυτά που περιμένουμε δεν τηρούνται από τις αρχές και τους άλλους ενδιαφερομένους. Εάν ε, λοιπόν δεν δούμε συγκεκριμένη δράση, θα πρέπει να αναλάβουμε άλλα βήματα και θα πρέπει να εξετάσουμε το όλο πλαίσιο των, ε, του προτιμησιακού καθεστώτος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κάριμ. Θα είμαι πολύ σύντομος. Σας ευχαριστώ για όλες τις παρατηρήσεις σας. Δύο θέματα θα ήθελα να θίξω πολύ σύντομα. Όταν συνομιλεί κανείς ε, με ε, παρασκευαστές ενδυμάτων στον Παγκλαντές, το βασικό επιχείρημα τους είναι αυτό που μόλις παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι οι τιμές των διανομέων σας είναι τόσο ανταγωνιστικές που διαβρώνουν το περιθώριο που χρειαζόμαστε για να ε, τηρήσουμε όλα αυτά που ζητάτε. αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση σε περιορισμένο βαθμό μπορεί να παρέμβει στη διαμόρφωση των τιμών. Υπάρχουν όμως κάποια πράγματα που μπορούμε να κάνουμε και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να τα κάνουμε. Επίσης υπάρχει το θέμα των ε, κατασκευαστών και της πρόσβασής τους στη χρηματοδότηση που χρειάζονται. Δεν ξέρω αν έχουν εκφράσει τις ανησυχίες τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε μένα πάντως σίγουρα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τις παρατηρήσεις τους. Νομίζω ότι πιο εύκολα θα μπορούσα να το συνοψίσω ως εξής. Μου θύμιζε τις ε, εκθέσεις στο σχολείο όπου μου έλεγε ο δάσκαλος ότι ο Καρίν τα πήγε πολύ καλά, μπορεί όμως να κάνει ακόμα περισσότερα. Ε, θα ε, κρατήσω λοιπόν, σημειώνω τις παρατηρήσεις σας ε, και θα δω τι μπορώ να βελτιώσω. Ε, πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Δεν μπορώ να πιστεύω ότι λέγανε τέτοια πράγματα για τις εκθέσεις σας στο σχολείο. Θα ψηφίσουμε την προφορική ερώτηση αύριο και η ε, προθεσμία για το ψήφισμα είναι Παρασκευή 5 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι και φτάνουμε στο τελευταίο θέμα της ημερησίας διάταξης. 20 λεπτά έχουμε στη διάθεσή μας και έχουμε δύο προσκεκλημένους. Παρακαλώ λοιπόν να τηρήσετε το χρόνο ομιλία σας. Είναι μια πολύ απλή ερώτηση. Θα πρέπει να χορηγηθεί στη ε, Σρι Λάνκα το σίγμα γάμα συν ε, δύο προς και κλειμένους έχουμε τον ε, κύριο Αλανκίναν ε, που ε, είναι αναλυτής και έχουμε και τον πρεσβευτή της Σρι Λάγκα, τον κύριο Ότνη Φερέιρα. Δίνω λοιπόν πρώτα το λόγο. Ε, Έλεν Κίναν, πέντε λεπτά παρακαλώ. Τος μικροφόνου. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Με μεγάλη μου χαρά και τιμή βρίσκομαι εδώ. Πέντε λεπτά δεν είναι πολύ χρόνο. Δεν θα προλάβω να πω όσα ήθελα να πω. Θα προσπαθήσω να είμαι περιεκτικό. Ε, ε, το δημοκρατικό άνοιγμα το 2015 της Σρι Λάνκα φώτισε την ε, παγκόσμια πολιτική σκηνή όπου υπονομεύεται η δημοκρατία. Η κυβέρνηση Εθνική Ενότητα της Σρι έγινε αποδεκτή από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υποσχέθηκε πολλές μεταρρυθμίσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σύσταση τον Ιανουάριο να χορηγηθεί ε, ε, ε, σίγμα γαμαπίσιν στη Σρι Λάνκα σύμφωνα με το αίτημά της. Ωστόσο, η Κομισιόν ήταν γενναιόδορη λέγοντας ότι δεν υπήρχε καμία έλλειψη εφαρμογής των διαφόρων ε, συμφωνιών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχουν γίνει και θετικές ε, αλλαγές, αλλά ακόμα δεν έχουν θεσμοθετηθεί και εξαρτώνται από την καλή βούληση των ηγετών της. Είναι πολλές οι ελλείψεις που αναφέρονται σε πρόσφατες εκθέσεις της, ε, είπα, της αρμοστίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ειδικών εισηγητών. Υπάρχει απόλυτη ατιμορρησία για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ε, πλήττει τη Σρελάνκα εδώ και δεκαετίες. Δεν έχει αλλάξει αυτό. Τώρα η επανεκκίνηση της διαδικασίας ε, ε, συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων δεν έχει αλλάξει στην πορεία. Ουσιαστικά επικεντρώνεται σε δύο βασικά ελλείμματα που σημειώνονται στην αξιόλογηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατά τα είναι θετική. Ε, και που είναι η μη συμμόρφωση με τη Διεθνή Συμφωνία ε, ε, Αστικών Δικαιωμάτων και την Συμφωνία κατά των βασανιστήριων. Έχει υποσχεθεί η Σρι να εφαρμόσει αυτές τις συνθήκες και η μεταρρύθμιση του ποινικού κώδικα ώστε οι κρατούμενοι να έχουν δικαίωμα ε, ε, αρρωγής από δικηγόρο. Ενώ φαίνεται ότι το Συμβούλιο και η Κομισιόν θα δώσουν το πράσινο φως ε, για το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων, οι μεταρρυθμίσεις αυτές δεν έχουν επιτευχθεί. Όσον αφορά την κατάρξη της PTA, η τελευταία έκδοση της νομοθεσίας κατά της τρομοκρατίας που θέλει να περάσει η κυβέρνηση ε, για να αντικαταστήσει την PTA υποβλήθηκε στην κυβέρνηση πριν λίγες μέρες ε, πριν από την ψηφοφορία την περασμένη εβδομάδα στο Κοινοβούλιο αυτή ε, η νομοθεσία περιλαμβάνει προβλήματα είναι πολύ ευρύς ο ορισμός του τρομοκρατίας υπενθυμίζει τις ρήτρε της PTA για τη σύλληψη των αντιφρονούντων ποινικοποιεί ε, τη συλλογή εμπιστευτικών πληροφοριών ε, και τελικά η πρόσβαση σε, ε, δικαστική, σε συνδρομή δικηγόρου εξαρτάται από κάποιες ρήτρε. Μια έκδοση έχει ήδη εγκριθεί από την κυβέρνηση σε μια ταχύα ψηφοφορία την περασμένη εβδομάδα, αλλά που περιλαμβάνει βάσει ενός αντιτύπου που ε, δημοσιεύτηκε σε μια ιστοσελίδα την περασμένη εβδομάδα ε, περιλαμβάνει δύο βασικά προβλήματα. Δεν λαμβάνει υπόψη ζητήματα σημαντικά που έχει επικρίνει η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωματών της Ριλανκά πριν από ένα μήνα βάσει ενός παλιότερου σχεδίου. Το νέο σχέδιο επιτρέψει αστυνομικού αστυνομικούς να απαγορεύσουν την πρόσβαση σε δικηγόρα εάν θεωρούν ότι μπορεί αυτό να επηρεάσει την έρευνα και ε, επίσης ε, περιλαμβάνει μια επικίνδυνη ρήτρα ε, για τη διαδικασία παρουσία δικηγόρου. Αυτά δεν φαίνονται πολύ σημαντικά σε ένα λιγότερο καταχρηστικό σύστημα και αφήνει ελεύθερα τα χέρια αστυνόμων και δικαστών και δικηγόρων. Για όλα αυτά τα ζητήματα δεν έχει επιτευχθεί ακόμα τίποτα. Και αυτά, ξέρετε, είναι μόνο νομοσχέδια. Το Κοινοβούλιο δεν έχει ακόμα ε, προχωρήσει με αυτά τα νομοσχέδια. Τα δύο αυτά βασικά ζητήματα δεν τα έχει λάβει επαρκώς υπόψη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξακολουθεί να υπάρχει η κράτηση πολλών ανθρώπων δυνάμει της PTA, δεν λειτουργεί η προστασία των θυμάτων, ε, ε απουσία διώξεων σε κάποιες περιπτώσεις. Ε, που έχει επισημάνει και το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών και δεν λειτουργεί το γραφείο των ε, αγνοωμένων. Αυτό δημιουργεί ε, προβλήματα στη διαδικασία που ζημιώνει την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαδικασία σύνταξης νέας ε, νομοθεσίας γίνεται με κλειστές πόρτες και, δεν επιτρέπ, και υπάρχουν κάποιες διαρροές σε εφημερίδες και έτσι γίνονται γνωστές οι προτινόμενες νέες νομοθεσίες στον ΟΗΕ. Παρότι ο ΟΗΕ ε, έχει δώσει τη σχετική επιτροπή την εντολή να συμβουλεύει την κυβέρνηση σε θέματα προστασίας των ανθρωπινών δικαιωμάτων. Καμία της νομοθεσίας ε, δεν έχει κοινοποιηθεί επίσημα στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το θέμα το νομοσχέδιο έχει κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρείται ως παροχή πληροφοριών σε ξένη κυβέρνηση. Πιστεύω λοιπόν ότι η διαδικασία αυτή ε, αν συνεχιστεί και χορηγηθεί το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων ε, θα απαιτηθεί μια αυστηρή διαδικασία παρακολούθησης αλλά θα είναι κάτι δύσκολο. Όπως μου είπε ένα ε, δημοσιογράφος, καθώς ερχόμουν στην συνεδρίαση αυτή, αφού χορηγηθεί η ΣΥΓΜΑ τι θα υποχρεώσει αυτού του ανθρώπου, την κυβέρνηση τη Ριλάγκα να υλοποιήσει την νομοθεσία που πρότεινε. Θα είναι νομική η μάχη. Έχω κάποιες προτάσεις, αν θέλετε να τις ακούσετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομος. Ευχαριστούμε για την κατανόηση που δείχνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, λέει ο πρέσβης. Μετά τις εκλογές του 2015, υπό την ηγεσία του Πρέδου και του Πρωθυπουργού, υποσχεθήκαμε στο λαό του Σιλάνκα ότι θα αλλάξει η κατάσταση της απομόνωσης για παράδειγμα και της αδικίας και θα συμπεριλάβουμε όλους τους εταίρους, φίλους και εταίρους προκειμένου να στηρίξουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα στον νόμο και να μην υπάρχει ατιμωρησία, για να υπάρχει χρηστή διακυβέρνηση υπέρ της ευημερίας του λαού μας. Η διεθνής κοινότητα πριν από μερικές εβδομάδες στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Γενέβη έκανε ένα σημαντικό βήμα προς τα μπρος με το ψήφισμα 30 καθετός 1 για μια παράταση δύο χρόνια παραπάνω. Και οι συζητήσεις προχωρούν ακριβώς για τη συμφιλίωση, για τη χρηστή διακυβέρνηση, για την ειρήνη και την οικονομική ευημερία όλων στη χώρα. Με ικανοποίηση διαπιστώνουμε ότι και 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταποκρίθηκαν στο ψήφισμα αυτό. Τα τελευταία δύο χρόνια η συνεργασία μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύθηκε. Τώρα έχουμε αξιωματούχο που συμμετέχει στις συναντήσεις μας, ομάδες εργασίας που ασχολούνται με την αναπτυξιακή συνεργασία, τις οικονομικές σχέσεις, την επανεισδοχή, τη διακυβέρνηση, το κρατοσδικαίο και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πριν από δύο χρόνια φτιάχτηκε σχετική ομάδα εργασίας. Επίσης υπάρχουν και αποστολές που ελέγχουν την κατάσταση όσον αφορά ε, την οικονομική ανάπτυξη και τη δημοκρατία στη χώρα. Υπήρξαν πολλές επισκέψεις στη χώρα τον τελευταίο χρόνο και με την αντιπροσωπεία για την Νότιο-Ανατολική Ασία και ήταν η πρώτη φορά εδώ και 10 χρόνια. Η συνεργασία μα επίση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενισχύθηκε ακόμα περισσότερο την προηγούμενη εβδομάδα, όπου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φιλοξένησε 10 βουλευτέ από την Σρι Λάνκα σε μια προσπάθεια να ενισχυθούν οι σχέσεις των δύο πλευρών. Πολύ σημαντικά όλα αυτά. Οι σχέσεις μας δηλαδή με τα Ηνωμένα Έθνη, την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες φιλικές χώρες για να ενισχυθεί δικιά μας πολιτική ανοίγματο σε συνεργασία με όλους τους εταίρους. Υπογραμμίζει επίσης και τη δικιά μας πεποίθηση ότι μια τέτοια συνεργασία θα είναι θετική για ε, την επίτευξη των στόχων της κυβέρνησής μας υπέρ της αηφόρου ανάπτυξης και της ε, βιώσιμης οικονομίας. Πολλά έχουν γίνει μέχρι τώρα, αλλά παραμένουν πολλά ακόμα. Ενίσχυση των θεσμών, ε, μεταρρυθμίσεις και οικονομική πρόοδος. Ε, ακούει όλες τις πλευρές η κυβέρνηση, μελετάει τα πράγματα, ανταλλάσσει πληροφορίες, παρακολουθεί τα σχόλια και επικοδομητικά δουλεύει με τους εταίρους για να αναλυθούν τα επόμενα βήματα που θα ασφαλίσουν ότι η Σρι Λάνκα θα είναι μια χώρα ευημερούσα που θα τηρεί την ποικιλομορφία και το κράτος δικαίου. Οι συστάσεις και παρατηρήσεις που γίνονται είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για μας. Στο στάδιο τώρα μετά τη σύγκρουση, διαπιστώσαμε πρώτα. Η κυβέρνηση αναλαμβάνει τις ευθύνες της όσον αφορά τις ανάγκες των ειδικών ομάδων που βγήκαν σημειωμένες από τον, τη σύγκρουση αυτή. Και αυτό με τη βοήθεια των εταίρων μας, μεταξύ άλλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια εθνική επίσης πολιτική για μια βιώσιμη λύση για την ε, ε, μετατόπιση του πληθυσμού γίνεται σε διαβούλευση με διάφορα υπουργεία αλλά και αρχές τοπικές και περιφερειακές και μη κυβερνητικές οργανώσεις. Επίσης θέλουμε να ακολουθήσουμε τους στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη του ΟΗΕ ώστε να υπάρξει μια οικονομική πρόοδος με τη συμμετοχή όλων. Το 2017 είναι το έτος ε, της ανακούφισης από τη φτώχεια στη Σρι Λάνκα με διάφορες εκδηλώσεις που έχουν οργανωθεί από ειδικού σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών. Θέλουμε την ειρήνη και τη σταθερότητα. Θα συνεχίσουμε να παίρνουμε μέτρα προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση στη χώρα σε συνεργασία με τους εταίρους μας υπέρ της χρηστής διακυβέρνησης θέλουμε δικαιώματα για όλους τους πολίτες σε μια δημοκρατική και ελεύθερη χώρα. Έχουμε δεσμευτεί υπέρ των ε, στόχων ε, της χιλιετίας επίσης, αναγνωρίζοντας τις επιπτώσεις που έχουν οι συγκρούσεις πάνω σε όλους τους πολίτες και θέλουμε να βοηθήσουμε για την ισότητα μεταξύ όλων και μεταξύ των δύο φύλων. Συνεργαζόμαστε με τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης με επικοδομητικό πνεύμα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για τη συμφιλίωση στη χώρα και για την ετήρηση και σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και περιμένουμε από αυτό να στηρίξει την Σρι Λάνκα για να αντιμετωπίσει τους τόσο δύσκολους στόχους που έχουμε μπροστά μας και κυρίως το στόχο της συμφιλίωσης. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ένα λεπτό κάθε συνάδελφος. Κυρία Καρίν, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, πιθανότητα να ξεπεράσω λίγο το χρόνο, διότι ο συνάδελφος Κρίστοφερ Φιέλνερ μου ζήτησε να μιλήσω ε, στο όνομά του. Αν μου επιτρέψετε λοιπόν μισό λεπτό παραπάνω, ε, ε, θα σας είμαι υπόχρεος. Συνάδελφοι, πρέπει να φροντίσουμε να μην μετακινούμε συνεχώς τον στόχο και τα ενιαία κριτήρια να ισχύουν και για την Σρι Λάγκα. Στις 11 Ιανουαρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ε, την αποκατάσταση του συστήματος ε, γενικευμένων προτιμήσεων για την Σρι Λάγκα, διότι ε, πληρεί τα κριτήρια όσον αφορά την τροτότητα και τις διεθνείς συμβάσεις, αλλά έχει λύσει και τις εκκρεμότητες που είχε επισημάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά την, αφαίρεση, την προηγούμενη αφαίρεση του καθεστώτος ΣΥΓΜΑΓΑΜΑΠΗ. Είχαμε πολύ σαφή ψηφοφορία την προηγούμενη εβδομάδα στην ε, Ολομέλεια και η κυβέρνηση της Σρι Λάγκα έχει εγκρίνει νέα συμφωνία πλαίσιο ε, σχετικά με τον ε, αντιτρομοκρατικό νόμο που θα αντικαταστήσει τον προηγούμενο, την προηγούμενη νομοθεσία. Θα ήθελα να ρωτήσω εάν θα μπορούσαμε να έχουμε περαιτέρω διευθυνήσεις σχετικά με το ακριβές χρονοδιάγραμμα σχετικά με τις τροπολογίες. Ίσως ο πρέσβης να μπορεί να μας διαφωτίσει. Από ό,τι καταλαβαίνουμε όμως ε, το νέο σχέδιο της νομοθεσίας ευθυγραμμίζει τον ε, αντιτρομοκρατικό νόμο με αυτά που αναγνωρίζονται διεθνώς σε επίπεδο ΟΗΕ η νέα ε, νομοθετική πράξη για τις ε, ποινικέ ε, διαδικασίες επίσης ευθυγραμμίζεται. Αυτά λοιπόν είναι τα συμπεράσματα της έκθεσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα που δημοσιεύθηκε φέτος και δείχνει τη δέσμευση της Φιλάνκα να συμμορφώνεται με τις διεθνείς της υποχρεώσεις. Οι μεταρρυθμίσεις βρίσκονται ψηλά στο θεματολόγιο αλλά δεν υπάρχει πάντα συμφωνία εντός της ε, κυβέρνηση συνασπισμού, το οποίο οδηγεί σε ε, καθυστερήσεις. Στις 11 ε, Μαΐου θα συζητηθεί το θέμα αυτό και θα έχει έτσι την ευκαιρία η κυβέρνηση της Ιλάνκα να υιοθετήσει απόφαση, αλλά είναι κάπως απίθανο να ξεφύγει από την θέση του Κοινοβουλίου στο θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Έξι λεπτά έχουμε στη διάθεσή μας, ε, δεν θα έχουμε μετά ε, του διερμηνεί στη διάθεσή μας, λέει ο ε, Αυτή λοιπόν είναι η πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε. David Μάρτιν, θα είμαι σύντομο. Θα ήθελα να καταστήσω σαφές ότι το SND συνεχίζει να πιστεύει ότι οι ελλείψεις όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου στη Σρι Λάγκα είναι ακόμα προφανής. Την προηγούμενη εβδομάδα αποφασίσαμε να αναγνωρίσουμε τα βήματα ε, της κυβέρνησης ε, παρά τις ε, ελλείψεις. Προτιμήσαμε λοιπόν να δούμε το ποτήρι ως μισογεμάτο αντί για μισοάδιο. Πιστεύουμε ότι έχουμε τώρα μια αφετηρία για περισσότερη εις βάθος συνεργασία και δεν θα πρέπει να θεωρηθούν όλα αυτά ούτε λευκή επιταγή ούτε το τέρμα. Και γι' αυτό θα ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την πρόοδο της Σρι Λάγκα. και θα θέλαμε να ακούσουμε ιδέες σχετικά με το πώς μπορεί να ενισχυθεί αυτή η συνεργασία. Επίσης, ε, η συνάδελφος που εκπροσωπώ θα ήθελε να ε, πει ότι είμαστε διατεθειμένοι να ξαναναστείλουμε την συμφωνία εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ εκπροσωπώ εδώ τη Λόλα Σάντσε, τη συνάδελφο που δυστυχώ δεν μπορούσε να είναι. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την προηγούμενη εβδομάδα ψήφισε ψήφισμα. Ε, το κατα... ψήφισε ουσιαστικά, το οποίο είχαμε υποβάλει συνάδελφο Λόλα Σάντσε και εγώ, που αναφερόμασταν στι συνθήκε που επικρατούν στην χώρα αυτή. Δυστυχώ παραμένουν πολλά προβλήματα στην χώρα. Μερικά από αυτά τα ακούσαμε ήδη. Πριν από μερικές εβδομάδες, τον Απρίλιο, με την Λόλα Σάντσεφ πήγαμε στην Σιλάνκα και συστήσαμε και με συνδικάτα και με εργαζόμενους και με την κυβέρνηση αλλά και με, κυ... με μη κυβερνητικές οργανώσεις και διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές παραβιάσεις και παραβιάσεις όσον αφορά τα εργασιακά δικαιώματα. Υπάρχει επίσης και η έκθεση του ΟΗΕ που αναφέρεται σε εκφοβισμό συνδικαλιστών, σε καταχρήσεις που γίνονται, σε εκφοβισμό από πλευράς της αστυνομίας και επίσης και σε βάρος των Ταμίλ πάνω απ' όλα. Θα είμαι σύντομος πρόεδρε, αλλά βλέπετε δεν μπορεί να παραβλέπουμε όλα αυτά τα πράγματα. Ποζεί ο λαός στη Σρι Λάγκα που φοβάται ότι θα χάσει τη δουλειά του ο κόσμος. Τα δικαιώματα των συνδικαλιστών πρέπει να γίνονται αποδεκτά, να υπάρχουν έλεγχοι και τα συνδικάτα και συνδικαλιστές να μπορούν να έχουν πρόσβαση στη δικαιοσύνη χωρίς εκφοβισμό. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας κάθε φορά που μιλάμε και για επενδύσεις. Και θα ήθελα να ακούσω από τον πρέσβη και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι θα κάνουν γι' αυτό. Τι θα κάνουν για να βελτιωθεί ο τρόπος με τον οποίο αναφέρεται η κατάσταση που επικρατεί στη χώρα εδώ. Ευχαριστώ. Είμαι μέλο τη Υποεπιτροπή Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και θα ήθελα να ακούσω και εγώ συστάσει για την παρακολούθηση εκεί. Από ό,τι καταλαβαίνω, η Γενική Διεθνήση Εμπορίου πρόκειται να συντάξει, έχει ήδη συντάξει έναν κατάλογο τον οποίο έχουν κοινοποιήσει στην κυβέρνηση της Σριλάνκα για συγκεκριμένα ζητήματα όπου χρειάζονται βελτιώσεις. Μπορούμε να έχουμε και εμείς ένα τέτοιο κατάλογο όπου να μπορέσουμε να προσθέσουμε κάποια θέματα. Ε, το ζήτημα, για παράδειγμα, των, δικαιωμάτων, ε, των έγκυων δικαιωμάτων ε, για αγιές που έχει καταλαβεί στρατός, για παράδειγμα. Ευχαριστούμε πολύ, η κυρία Λάμπερτς. Ευχαριστώ Μιλώ ω πρόεδρος της Αντιπροσωπείας για την Νοτιά Ασία. Πολλοί από εμά αισθανόμαστε απογοήτευση. Δεν υπάρχει απτή πρόοδος, όπως είδαμε. Πολλά λόγια, αλλά λίγα έχουν ε, γίνει νομοθεσία μετά τη νέα κυβέρνηση. Εκεί υπάρχουν προβλήματα. ενώ η κοινωνία των πολιτών ελπίζει πραγματικά ότι θα μπορούσαν να γίνουν αλλαγές και ότι θα πρέπει να γίνουν. Και στη δική μου πολιτική ομάδα συμμεριζόμαστε πολλές από τις ανησυχίες του David Μάρτιν. Πρέπει να δούμε σοβαρά πώς θα πραγματοποιήσουμε την παρακολούθηση και πώς θα συμμετέχει σε αυτήν η κοινωνία των πολιτών ώστε και αυτή να αποτελέσει κομμάτι της λύσης ε, στο πλαίσιο ορισμένων ε, συμφωνίων όπως η CCPR. Και ο τρόπος που θα αντιμετωπίσει το όλο θέμα Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποτελέσει επίσης κομμάτι της λύσης που θέλουμε να δούμε στη Σρι Λάνκα. Ευχαριστούμε ένα λεπτό για τον κύριο Κίναν για να μας δώσει τις ιδέες παρακολούθησης και μισό λεπτό για την Κομισιόν να απαντήσει την ερώτηση. Της κυρίας Λόπουλα. Κυρία Μπεγκέν, θέλετε να πείτε κάτι. Ωραία, ένα λεπτό. Ε, ευχαριστώ πρόεδρε. για την παραχώρηση αυτού του προτιμησιακού συστήματος. Εμείς είμαστε υπέρ του να βοηθάμε τις φτωχότερες χώρες. Αλλά στη χώρα αυτή, όπου υπήρξε αυτός ο μεγάλος ε, ε, ε, πόλεμος με παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που σύμφωνα με τον ΟΗΕ μόνο τους τελευταίους μήνες οδήγησε σε 40.000 νεκρούς και παραπάνω, εμείς θα θέλαμε να υπάρξουν κάποιες αμφιβολίες, λίγο πιο έντονες. Για τον λόγο αυτό, εμείς θα προτιμούσαμε να είχαμε περισσότερο χρόνο για να λάβουμε περισσότερες εγγύησεις, καλύτερα αποτελέσματα, για να γίνει κάτι με αυτές τις ε, ε, ε ε, που κατασχέθηκαν ε, να γίνει κάτι με το όργανο αναζήτησης των αγνωμένων πολέμου και για να επιτευχθεί κάποια ε, συμβιβασμός. Ξέρουμε ότι ασκούν πολλές πίεσεις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να πάνε στη Στριλάνκα να παράγουν με, σε χαμηλές τιμές με τοπικούς εργαζομένους, αλλά το θέμα εδώ δεν είναι να το ότι είναι μισογεμάτο ή μισοάδιο. Το θέμα είναι να έχουμε ένα όπλο που θα μας ωφελήσει. Και Εμεί, ε, η συνείδησή μα, δεν μας επέτρεψε να ψηφίσουμε κάτι τέτοιο. Ε, ευχαριστούμε κύριο Σκέναν. Έχετε ένα λεπτό. Συμβουλές για την παρακολούθηση. Ευχαριστώ πολύ. Η ομάδα μας ε, θα δημοσιεύσει σύντομα έκθεση που θα παρουσιάζει πιο αναλυτικά το θέμα αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εργάζεται με πιο συστηματικό τρόπο, να ε, συνεργάζεται με το γραφείο του ΥΠΑ του Αρμοστή για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εκεί υπάρχουν πολύ ικανοί άνθρωποι. περισσότερη συνεργασία λοιπόν. Πιστεύω όμως επίσης ότι θα πρέπει να ενισχύσει την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Σρι Λάγκα. Η Σρι Λάγκα δεν έχει τηρήσει τις υποχρεώσεις της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της θα πρέπει να πιέζει την κυβέρνηση της Σρι Λάγκα να αυξήσει το δυναμικό αυτής της Επιτροπής ε, και να επιτρέψει στην Επιτροπή αυτή να ε, κάνει τη δουλειά της ε, και να διευρύνει τις ε, αρμοδιότητές της. Κάθε... Πιστεύω επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να χρηματοδοτήσει την Επιτροπή αυτή για να την ενισχύσει ιδιαίτερα τα περιφερειακά της γραφεία που έχουν παίξει θετικό ρόλο και έτσι μπορούν να αποτελέσουν δίοδο για την συνεργασία και την επικοινωνία με την κοινωνία των πολιτών. Σας ευχαριστώ πολύ για την ε, σύντομη απάντησή σας. Ε, αργότερα θα ακούσουμε περισσότερες λεπτομέρειες δηλαδή από εσά και τι γίνεται σχετικά με τον κατάλογο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, μπορεί να τεθεί στη διάθεσή μας να σας απαντήσω κατευθείαν είναι κατάλογος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης για τα ανθρωπίνα δικαιώματα. Δεν είναι δικός μας κατάλογος για το σύστημα ΣΥΓΜΑΓΑΜΑΠΗ θα στείλουμε επιστολή όπως στέλνουμε σε όλους τους δικαιούχους. Ε, δεν έχει γίνει αυτό όμως στο πλαίσιο του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων. Εμεί δεν έχουμε κατάλογο. Φαντάζομαι ότι αναφέρεστε σε αυτόν τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση. Ωραία, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούσαμε λοιπόν τι ε, συμβουλέ, ακούσατε μάλλον τι συμβουλέ ε, για ε, τη διαδικασία παρακολούθηση. Σα ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρέσβη. Αξιότιμη προσκεκλημένη για τη συζήτηση αυτή. Έτσι, ολοκληρώνουμε την συζήτησή μα για το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων στη Σρι Λάγκα. Ε, θα τα πούμε αύριο στι 9 η ώρα.